So, schönen guten Morgen. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω όλους. Ναι, κουκού. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω στην τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις διακοπές. Έχουμε σήμερα υψηλούς προσκεκλημένους από την Εστονία. Καλωσορίζω τον κύριο Γευγένη Οσινόφσκι, Υπουργό Εργασίας και Υγείας. Και την συνάδελφό του, την κυρία Κάια Ήβα, την Υπουργό Κοινωνικής Προστασίας. Έχουμε μέχρι τις 10.30 ακριβώς ε, τα θέματα μας. Ε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια παρουσίαση της κυρίας Υπουργού και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Οσινόφσκι. Ε, αν τα καταφέρετε σε πέντε λεπτά θα είναι καλά, αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε χρόνο για να επεκταθούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίδετε να παρουσιάσω τα σχέδια και προτεραιότητες της Εστονικής ε, Προεδρίας. Η κοινωνική προστασία, η κοινωνική ασφάλιση, πολιτική για τα παιδιά και για την οικογένεια εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου και θα αναφερθώ στις προτεραιότητες μας αυτούς τους τομείς και ο κ. Σινόφσκι θα αναφερθεί στους δικούς του τομείς. Η Εσθονία έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για πρώτη φορά και σύνθημά μας για αυτή την Προεδρία είναι ενότητα μέσω ισορροπίας. Ο βασικός στόχος σαν χώρα που έχει την Προεδρία είναι να κρατήσουμε την Ευρώπη ενωμένη προσπαθώντας να πετύχουμε ισορροπίες μεταξύ διαφόρων κομμάτων, ιδεών, αξιών και πράξεων. Στον τομέα των κοινωνικών θεμάτων θα θέλαμε η Ευρώπη να είναι μια ενωμένη ένωση που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες κάθε πολίτη και αυτό βάσει κοινών αξιών όπου κάθε άνθρωπος έχει ζωτική σημασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό τώρα, διότι η πίστη των ανθρώπων στην προστιθέμενη αξία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρχίσει να κλονίζεται. Γι' αυτό οι θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελεύθερη διακίνηση ατόμων και οι ίσες ευκαιρίες είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να τα εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια από τις προτεραιότητες της Εσθονίας είναι να υποστηρίξει την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Αν δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι ή να εγκατασταθούν σε κάποια άλλη χώρα, αν δεν μπορούν να ωφεληθούν από διάφορα κοινωνικά επιδόματα, τότε δεν υπάρχει εγγύηση για την ελεύθερη διακίνηση. Γι' αυτό βασική νομοθεσία για μας συμπεριλαμβάνει και την επικαιροποιημένη, το επικαιροποιημένο κανονισμό για το συντονισμό των κοινωνικών μέτρων. στα κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών έχουν αλλάξει οι περιστάσεις και πρέπει οι κανόνες να γίνουν διαφενέστεροι, πιο εύληπτοι και να είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν. Βασιζόμαστε στη δουλειά που έχει κάνει η Μάλτα, ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο πάνω σε δύο δύσκολα θέματα, την ίση αντιμετώπιση όσον αφορά την πρόσβαση στα ευεργετήματα και ε, το εφαρμοστείο δίκαιο. Αυτά είναι περιπλοκότατα θέματα και πάρα πολύ ευαίσθητα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μια ε, συμφωνία στο τέλος που θα είναι σαφής και δίκαιη. Οι Μαλτέζοι συνάδελφοι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και θέλουμε να συνεχίσουμε επί προεδρίας μας ανοίγοντας δύο κεφάλαια μακροπρόθεσμη μέρημνα και τα διάφορα οικογενειακά επιδόματα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θέλουμε να καταλήξω συμφωνία στο Συμβούλιο όσον αφορά αυτά τα τέσσερα ζητήματα που σας ανέφερα. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι κανόνες είναι εύληπτοι για τον κόσμο και διαφανείς. Και αυτό πρέπει να αντικατοπτήσει στα κείμενά μας. Συνάδελφοι, η Ευρώπη ποτέ δεν θα καλύπτει τους πάντες εάν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα δικαιώματα όλων ε, παρά τις διαφορές τους με μια γυράσκουσα κοινωνία είναι επιτακτική ανάγκη να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες. Όχι αφηρημένα. Τα δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν μια αφηρημένη υπόσταση, πρέπει να βρούμε πρακτικές λύσεις όπως το θέμα της οδηγίας της προσβασιμότητας. Στόχος μας εκεί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστεί σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Γνωρίζουμε ότι η οδηγία προσβασιμότητας θα μας ε, οδηγήσει σε δύσκολες συζητήσεις. Από τη μια πλευρά πρέπει να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να ζουν ανεξάρτητοι και να μπορούν ε, να συμμετέχουν στην κοινωνία και να λαμβάνουν ε, αποφάσεις με ανεξάρτητο τρόπο. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβάλλουμε κάτι παραπάνω από τις αναλογικές απαιτήσει ε, στις επιχειρήσεις και να προωθήσουμε την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτός ένας συμβιβασμός. Καλή βούληση και τιμότητα συνεργασίας από πλευράς κρατών μελών θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επ' αυτών στο Συμβούλιο στις 12 και στις 13 Οκτωβρίου στο Ταλίν θα γίνει διάσκεψη εμπειρογνωμόνων με θέμα τη μετάβαση από υπηρεσίες με θεσμική βάση σε υπηρεσίες με κοινωνική, κοινοτική βάση. Συγγνώμη. Και αυτό αφορά επίσης την ε, διαβίωση με ανεξάρτητο τρόπο, αν θέλουμε να ανταλλάξουμε βέλτιστες ε, πρακτικές, γνώσεις για λύσεις εφικτές που δίνουν αποτελέσματα, ούτω ώστε να μπορεί ο κόσμος να ζει αξιοπρεπώς και ανεξάρτητα. Το Συμβούλιο θα υθετήσει σχετικά συμπεράσματα. Εν κατακλείδη, να σας υπενθυμίσω ποιο είναι το σύνθημα της Προεδρίας μας. Ενότητα μέσω ισορροπίας είναι το σύνθημά μας. Συνάδελφοι, η εσθονική Προεδρία θα είναι επιτυχής ανάλογα με τη διάθεση συμβιβασμού των εταίρων μας. Ελπίζουμε η συνεργασία μας να είναι επικοδομητική και εύχομαι σε όλους μας μια πολύ επιτυχή εστονική προεδρία. Ευχαριστώ. ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, μετά τόσο είπε η συναδελφός μου, εγώ θα μιλήσω λίγο περισσότερο για τις προτεραιότητες που έχουμε στα θέματα τα κοινωνικά και της απασχόλησης. Όπως είπε ήδη η Υπουργός, η κυρία Ήβα, η κοινωνική Ευρώπη που θα στηρίζει την κινητικότητα της εργασίας είναι προτεραιότητα για την Προεδρία μας. Σκεφτόμαστε την κοινωνική Ευρώπη στο πλαίσιο της ψηφιακής κοινωνίας. Θεωρούμε ότι είναι προαπαιτούμενο για μια καινοτόμο και ψηφιακή Ευρώπη, που είναι άλλη μια οριζόντια προτεραιότητα για την Εστονική Προεδρία. Στο πεδίο της απασχόλησης εστιάζουμε στην κινητικότητα της εργασίας. Σκοπεύουμε να πετύχουμε συμφωνία στο Συμβούλιο για την οδηγία απόσπασης εργαζομένων. Θέλουμε να βρεθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ αφενός της διασφάλισης των αποσπασμένων εργαζομένων και αφετέρου της ελευθερίας των εταιριών να παρέχουν υπηρεσίες. Είναι ένα δύσκολο θέμα όπως καταλαβαίνουμε και αφορά ακριβώς ε, το ίδιο, την ίδια την καρδιά του ευρωπαϊκού ιδεώδους όπου έχουμε δύο αξίες την ε, ελεύθερη διακίνηση αλλά και την δικαιοσύνη από την άλλη πρέπει να ισορροπήσουν θα συνεχίσουμε την δουλειά των Μαλτέζων ε, συναδέλφων για να βρεθεί μια ισορροπία για να βρεθεί ένα συμβασμό που θα μας επιτρέπει να έχουμε ένα σαφές κείμενο το οποίο θα μπορεί και να εφαρμοστεί. Είμαστε φιλόδοξοι και θέλουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία στο Συμβούλιο μέχρι το Συμβούλιο του Οκτωβρίου και μετά ε, θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μαζί σας. Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, ε, η ψηφιοποίηση, έχει βαθύτατα αποτελέσματα στις ε, κοινωνίες μας. Και καλωσορίζουμε άρα την πρόταση της ε, Κομισιόν για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες μας για το τι εστί η Ευρώπη. Πολλά από αυτά τα δικαιώματα βεβαίως υπάρχουν ήδη στα περισσότερα κράτη-μέλη, κάποια άλλα όχι, αλλά το κυριότερο ο πυλώνας είναι μια πολιτική δέσμευση της Ένωσης που τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ε, βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ε, ίσες ευκαιρίες και επαρκή κοινωνική προστασία. Η επιθυμία μας είναι να προχωρήσουν οι συζητήσεις στο πολιτικό επίπεδο, στο Συμβούλιο, και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι εξίσου φιλόδοξο με μας και μαζί με την Κομισιό να μπορούμε να υπογράψουμε τη σχετική διακήρυξη μέχρι το τέλος του έτους για να εγγυηθούμε στις ευκαιρίες για όλους στην αγορά εργασίας θα πρέπει να προωθήσουμε τα μέτρα για την ισορροπία οικογενειακής και εργασιακής ζωής που θα προωθήσουν επίσης ε, το πώς θα μοιράζονται καλύτερα τις ευθύνες οι γονείς για να μπορούν και οι γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας και οι άντρες να συμμετέχουν στην οικογενειακή ζωή. Έτσι, θα συζητήσουμε ακριβώ το σχέδιο αυτό οδηγίας επιπλέον. Συγκεκριμένα σχέδια για αυτό το θέμα θα συζητηθούν και στο άτυπο συμβούλιο στο Ταλίν την επόμενη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του Ατυπού Συμβουλίου επίσης θα επικεντρωθούμε και στις νέες μορφές οικογένειας και εργασίας. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ποιότητα της εργασιακής ζωής και του εργασιακού περιβάλλοντος. Έχουμε τις ε, προτάσεις ε, για την οδηγία για τις καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες ε, επί τις οποίες θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκοπεύουμε να ε, συμβιβάσουμε τις αποκλίνουσες απόψεις. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στις αλλαγές ε, της οικονομίας και της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα στο συνέδριο για τις νέες μορφές εργασίας στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο Ταλίν που στόχο έχει να εξετάσει τις προκλήσεις και την κοινή μας αντίδραση. Με βάση αυτές τις συζητήσεις ε, θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου για το μέλλον της εργασίας. Γνωρίζουμε ότι εκπληρώνοντας όλα αυτά θα έχουμε την στήριξή σας και βεβαίω χρειάζεται καλή ανάλυση για να ασκήσουμε σωστή πολιτική. Γι' αυτό έχουμε και τις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας βοηθούν και τους σχετικούς κανονισμούς, τους συντηρητικούς κανονισμούς των υπηρεσιών αυτών. Αναμένουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους και καλωσορίζουμε την έμφαση που αποδίδεται σε κάθε μία από αυτές τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και αναμένουμε να προωθήσουμε το πακέτο μας. Όπως ξέρετε, η φύση και η ουσία του κειμένου είναι τα ίδια και βεβαίως απαιτείται και από σας η ευελιξία. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα έχουμε διάφορα θεμελιώδη και δύσκολα ζητήματα να αντιμετωπίσουμε όμως. Σας διαβεβαιώ ότι με την συνάδελφό μου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουδιέ. Στην Επιτροπή μας η διαδικασία έχει ως εξής. Πρώτα απ' όλα θα πάρουν το λόγο οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά σε μια δεύτερη διαδικασία ερωταποκρίσεων οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να σημειώσετε τις ερωτήσεις για να απαντήσετε κατόπιν αφού πάρουν το λόγο όλοι οι συνάδελφοι. Είναι απλούστερο αυτό. Πρώτος, ο συνάδελφος David Κάζα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την παρουσίασή σας. Η Προεδρία σας αρχίζει σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, μια περίοδο κατά την οποία Όλοι θέλουμε να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα για την αύξηση της απασχόλησης, για την εκπαίδευση, την ε, αντιστοίχηση δεξιοτήτων με τις θέσεις ε, εργασίας και την, με, κυκλοφορία των εργαζομένων. Στην Ευρώπη είμαστε περήφανοι που από τη μία έχουμε ισχυρές, σταθερές δημοκρατίες και τι ισχυρότερε προδιαγραφέ κοινωνική προστασία από την άλλη. Ας ελπίζουμε ότι θα παραμείνει γι' αυτό καλό την Προεδρία σα να προστατεύσει τι αξίε μα και τις ελευθερίες όπως ε, αναφέρονται στις συνθήκες η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας του ε, δικαίου εμπορίου και της αλληλεγγύης, οι αρχές όλες αυτές πρέπει να είναι η προμετωπίδα οποιονδήποτε συζητήσεων κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η Προεδρία σας έχει ως σύνθημα την ενότητα μέσω της ισορροπίας. Μ' αρέσει το σύνθημά σας. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να επιτύχει η Προεδρία σας ούτως ώστε να συμβαστούν οι διαφορές απόψεων για τα θέματα αυτά. Για παράδειγμα, η εχθρότητα προς την ε, ενιαία αγορά πρέπει να αντιμετωπιστεί για να αποκτήσει νέα ορμή η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Πρέπει να εστιάσετε όχι μόνο στα τεχνικά θέματα, αλλά και την πολιτική τους διάσταση για να επιτύχουμε τα περισσότερα για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Για τους σοσιαλιστές. Υποθέτω ότι θα πάρει το λόγο η Άγνε Γιονγκέριου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους Υπουργούς για τις ε, παρουσιάσει τους. Και εμένα μου αρέσει ο, ο, ο τίτλος, το σύνθημα της Προεδρίας σας. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα που όλοι θέλουμε να λύσουμε, πώς θα διατηρήσουμε την ενότητά μας, αλλά με ισορροπημένο τρόπο. Είναι βεβαίως η πρώτη προεδρία σας. Οπότε, καταρχάς, να σας συγχαρώ για τον μόλις επιτυχώς ε, τα διάλογο για τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Γιατί βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καλός ενός για την έναρξη της Προεδρίας σας το ότι τελείωσε ο τριμερής διάλογος για το πρώτο τμήμα αυτής της οδηγίας. Δεύτερον, όπως είπε και ο συνάδελφος Κάζα, είναι κρίσιμη η συγκύρια σε όλη τη διαδικασία της θητείας μας και της Επιτροπής. Τώρα πρέπει να επιτύχουμε αποτελέσματα για ορισμένα κοινωνικά θέματα. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τριπλό α για τα κοινωνικά θέματα. Πρέπει λοιπόν να το επιτύχουμε. Χάρηκα επίσης που σας άκουσα να λέτε ότι θέλετε να καταλήξει το Συμβούλιο για την Οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων στη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών για να μπορέσει να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος υπό την Προεδρία σας. Αυτό θα ήταν μεγάλη ανακούφιση για μένα, αν επιτευχθεί. Έχω μία ερώτηση. Που έχει να κάνει με τον τριμερή διάλογο για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και συγκεκριμένα του Σώματος Αλληλεγγύης. Βεβαίως, είναι θέμα που θα συζητήσετε. Είναι καλή αρχή να ξεκινήσουμε με το σώμα αλληλεγγύης. Αλλά αν δεν υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση για αυτό το εγχείρημα, Άρα τι θα γίνει. Θα πάρουμε από άλλα κοινωνικά προγράμματα τη χρηματοδότηση. Προγράμματα που μας ενδιαφέρουν και εσάς και εμάς πολύ. Άρα πώς θα επιτύχουμε τη σωστή ακριβώς ισορροπία μεταξύ του Σώματος Αλληλεγγύης και του Κοινωνικού Ταμείου και του Έρασμος ΣΥΝ. Ευχαριστώ. Ισιά τώρα. Ανθία Μάκιντάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργή, κυρία και κύριε Υπουργέ. Πολύ καλή παρουσία εδώ. Και εγώ λοιπόν ε, χαιρετίζω το σύνθημα της Προεδρίας σας. Ενότητα μέσω αλληλεγγύης. Ε, μέσω ισορροπίας, συγγνώμη. Ιδιαίτερα για την ε, νομοθεσία, για την απασχόληση, είναι βασικό να επιδιώκουμε πάντα την ισορροπία. Χαιρετίζω λοιπόν την ιδέα σας ότι οι κανόνες πρέπει να είναι εύχριστοι. Εγώ ξέρετε παλιά ήμουν επικεφαλής μιας μικρής επιχείρησης και για τις μικρές επιχειρήσεις το ιδανικό είναι να μην χρειάζεται να κάνεις μεγάλη προσπάθεια για να ερμηνεύεις, να κατανοείς ή να χρειάζεσαι να πληρώσεις και ειδικού για να σου τις ερμηνεύσουν. Πρέπει λοιπόν να είναι εύχρηστοι κανόνες, να είναι εύκολο να τους καταλάβει και να τους εφαρμόσει μια μικρή επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι ζουν και ε, λειτουργούν σε καθεστώς ασφάλειας και δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να διαπιστώσουν ότι παρέβησαν τον νόμο χωρίς να το καταλάβουν. Και ένα από τα θέματα που αναφέρατε ιδιαίτερα είναι η απόσπαση των εργαζομένων. Εδώ λοιπόν θέλουμε κανόνες που να είναι εύκολο να γίνουν κατανοητοί και όπου θα πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητα των τόσο διαφορετικών χωρών στην Ευρώπη και των διαφορετικών ενδιαφέροντων και προοπτικών. Και είναι πολύ σημαντικό που θα αναλάβει η Εστονία τώρα την Προεδρία. Γιατί φοβάμαι ότι υπάρχει κίνδυνος διαφοροποιήσεων μεταξύ των νέων μικρότερων χωρών και των μεγάλων παλαιότερων όπου οι μισθοί είναι μάλλον υψηλότεροι στη Δυτική Ευρώπη δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί και η φωνή των νέων μικρότερων χωρών. Και θα ήθελα κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Πού βλέπετε την ισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ούτως ώστε να διατηρήσουμε την ενότητά μας, αλλά παράλληλα να καταλήξουμε σε μια οδηγία για την απόσπαση που να μας εξυπηρετεί όλους και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, Η Μαρτίνα Γκλαμπάιοβα. Ναι, ναι, ε, θα μιλήσω εγώ για να προλάβει ο συντονιστή μου να θέσει ερωτήσει στον επόμενο γύρο. Ευχαριστώ για τις, ε, τις παρουσιάσεις σας. Έχετε πολλές προκλήσεις. Και δεν είναι εύκολη η συγκυρία για την Ευρώπη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, αλλά καλά τα πάτε. Η φωνή σας ε, ήδη ακούγεται χάρη και στους συνεργάτες σας γιατί νομίζω ότι οι συνεργάτες σας ε, εργάζονται πολύ σκληρά, ήξεραν τις προτεραιότητες σας πολύ πριν ξεκινήσει η Προεδρία. Θα σας κάνω μια ερώτηση προς τον Υπουργό Σινόφσκι και έχει να κάνει όπως και προηγούμενη με την οδηγία για την απόσπαση. με μία από τις Κιώδης, από μία μικρή χώρα, από την Τσεχική Δημοκρατία. Χρειάζεται λοιπόν ε, ανάγκη, υπάρχει ανάγκη λοιπόν για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. Κύριε Υπουργέ, και εσείς αυτή τη στιγμή έχετε αποσπαστεί στις Βρυξέλλες. Ελπίζω να μην είχατε δυσκολίες ε, στα σύνορα του Βελγίου, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει πιο δύσκολη κατάσταση στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να την ε, αντιμετωπίσουμε. Είπατε ότι θέλετε να ακούσετε και τις δύο πλευρές. Θεωρώ ότι η Εστονία είναι πολύ καλό συντονιστή αυτή τη συζήτηση. Και αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση. Να καθίσετε στο τραπέζι και με τις δύο πλευρές και να καταλήξετε. Και βεβαίως θα ακούσετε και διαφορετικές προσεγγίσεις και στο Συμβούλιο. Ιδιαίτερα όπως είπε και η Υπουργό Ήβα, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να διατηρήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών και αυτούς θέλετε να στηρίξετε. Και σας εύχομαι καλή συνεργασία και με τους συναδέλφους των μεταφορών γιατί το πακέτο κινητικότητας έχει αυτές τις δύο πλευρές. Μία ερώτηση στην ε, κυρία Εύα για τον συντονισμό στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Συζητάμε πολύ για το ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος των πληρωμών και προς ποιους και τα λοιπά, των επιδομάτων δηλαδή, αλλά πρέπει να είναι και αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων των νομοθετημάτων που εγκρίνουμε. Μήπως θα μπορούσατε να προωθήσετε σε αυτό το κλάδο κάποιες ψηφιακές λύσεις. Ίσως κάποια ανταλλαγή στοιχείων για θέματα κοινωνικής ασφάλειας, ποιοι λαμβάνουν ποια επιδόματα για να καταπολεμηθούν οι απάτες. Θα ήταν πολύ καλό κάτι τέτοιο νομίζω. Γενικά ψηφιοποίηση ή καινοτομία. Αυτά δεν σταματάνε ποτέ και δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Ίσως η Εστονία θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα για πολλούς άλλους. Ίσως να προτείνει νέες λύσεις για τον κοινωνικό συντονισμό και την απασχόληση. Και σας ενθαρρύνω να ανταλλάξετε και να μοιραστείτε με εμά βέλτιστες πρακτικές, γιατί τα πάτε πολύ καλά σε πολλούς τομείς και το βλέπω καθημερινά. Γιατί έχω έναν καταπληκτικό εστονό σύμβουλο και νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ τη Τσεχική Δημοκρατία και τη Εστονία και η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Τα πάει πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρο για την ε, αριστερά. Η Παλώμα Λόπεθ Βερμέχων. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα ενημέρωσης από πρώτο χέρι επί των προτεραιοτήτων της Εστονία για το προσεχέ εξάμεινο. Κάποια σχόλια για τον κοινωνικό πυλώνα. Όλοι ξέρουμε ότι ο κοινωνικό πυλώνας είναι προ το παρόν ε, μεγαλοστομία χωρίς ε, νομική ε, υφή. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωριστούν τα κοινωνικά δικαιώματα που ανήκουν σε αυτόν τον κοινωνικό πυλώνα και θα πρέπει να μεταφραστούν σε ενωσιακή νομοθεσία. Ενωσιακή λέω. Γιατί αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ δεν εξυπηρετούν λύσεις δύο ταχυτήτων. Στα πλαίσια αυτά. Επιμένω να διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις. Για να εμβαθύνουμε. Να δούμε λοιπόν, εάν θέλετε να διερευνήσετε τις δυνατότητες ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως προβλέπουν οι συνθήκες, ή και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κάρτη, ε, Χάρτη, συγγνώμη, για να υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ των διαφόρων διεθνών συμβάσεων που καθορίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Και αναφέρομαι ακριβώ στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και θα ήθελα να ξέρω, διότι ένα θεμελιώδε στοιχείο αυτού του προτύπου είναι η σχέση που έχουν μεταξύ του οι κοινωνικοί εταίροι. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί κάποια πρωτοβουλία για να ενισχύσετε το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια ακριβώς Τη Ένωση, δηλαδή σε ενωσιακό επίπεδο. Τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο. Μιλήσατε για τη θέση σας για, για τους αποσπασμένους. Με ανησυχεί ότι θέλετε να επιτύχετε την ισορροπία μεταξύ της ενιαίας αγοράς και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ενώ η μεταρρύθμιση αυτής της οδηγίας θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση των εργασιακών κανόνων γιατί δυστυχώ αυτό δεν συμβαίνει. Αν μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα θα σας ήμουν ευγνώμων. Διότι έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα της μεταγραφής της οδηγίας, της εφαρμογής της οδηγίας, της απόσπασης. Που θα έπρεπε να έχει περάσει στις εθνικές νομοθεσίες, αλλά δεν συμβαίνει. Και ορισμένες χώρες Ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει ε, και διαδικασίες ε, επί παραλήψη για τη μην ε, μεταγραφή. Και τώρα... Ο για Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους Υπουργούς. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο κατά το εξάμεινο της Προεδρίας σας. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται προς τον Υπουργό Καγιαΐβα. Από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που είπατε, αναφερόσασταν σε παρόμοιο επίπεδο ε, χρηματοδότησης της στήριξης των διαφόρων μέτρων. Μπορείτε να είστε πιο ακριβείς όσον αφορά το θέμα αυτό. Μετά τη γενική προσέγγιση που θα ακολουθήσατε όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα για μια οικογένεια, για ένα νοικοκυριό. Τώρα επεξεργαζόμαστε το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το ελάχιστο εισόδημα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έδωσε μια πρόταση οδηγίας σχετικά με το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η θέση σας όσον αφορά αυτό το ελάχιστο εισόδημα, την ελάχιστη αμοιβή. Αναφερθήκατε στην απόσπαση των εργαζομένων και τη σχετική οδηγία. Αυτό σαφώς συνδέεται με το πρόβλημα αυτό της ελάχιστης αμοιβή και του ελάχιστου εισοδήματος. ελάχιστο ημερομίσθιο για τη Λετωνία είναι πέντε φορές μικρότερο ε, από το Λουξεμβούργο. Παρόμοιος ο συσχετισμός ε, μεταξύ Εσθονίας και Λουξεμβούργου όσον αφορά το ελάχιστο ημερομίσθιο. Χωρίς να λυθεί το πρόβλημα αυτό, δεν μπορούμε να λύσουμε και προβλήματα και αντιθέσεων αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Εφόσον ε, σύνθημά μας είναι ίση αμοιβή για ίση εργασία. Μπορούμε κάπου να προσθέσουμε ίση αμοιβή για ίση δουλειά οπουδήποτε. Εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Ε, οι πιο πλούσιες χώρες δίνουν πενταπλάσια αμοιβή από ότι οι φτωχότερες χώρες προς τον Υπουργό τον κύριο Σινόσκι. Η μελλοντική οδηγία που αφορά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής εξηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι προθέσεις της οδηγίας. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό ο τελικός απολογισμός, αλλά δημιουργήθηκαν και κάποια ερωτηματικά. Η διάρκεια της άδειας, της γονικής άδειας, είναι κάτι που μας απασχολεί και διότι η ισχύουσα οδηγία για τη γονική άδεια δεν έχει δώσει θετικά αποτελέσματα. Έχετε κάποια απάντηση να δώσετε σχετικά με αυτά μητρική ε, άδεια για τις μητέρες και ε, γονική άδεια. Σας ευχαριστώ. Για το EFTD δεν βλέπω κάποιον εδώ. Όχι, κανείς. Για το ENF επίσης δεν βλέπω κανέναν. Καλώς. Άρα κλείνουμε εδώ με τους συντονιστές και μπορούμε να περάσουμε στις απαντήσεις. Παρακαλώ. Ποιο θα ξεκινήσει. Κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, για την Προεδρία μας, που μόλις τώρα ξεκινάει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας ε, για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσω να δώσω τώρα κάποιες απαντήσεις. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι το γενικό ερώτημα του που αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και πώς θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που αφορούν ευαίσθητους τομείς και πώς θα πετύχουμε συμφωνίες σε ζητήματα όπως ο κανονισμός περί συντονισμού. Με τη Βουλγαρία και με την Αυστρία συνεργαστήκαμε πολύ καλά και όλοι μαζί θέλουμε να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα για το συντονισμό για την κοινωνική ασφάλιση, να έχουμε μια κοινή θέση μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2018. Ε, θέλουμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν όλες οι πλευρές, ούτως ώστε αυτά τα κείμενα να είναι εύληπτα, να ερμηνεύονται εύκολα και να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις όλων. Επίσης, θέλουμε να έχουμε ξεχωριστές νομικές βάσεις για να πετύχουμε σε κάθε χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όσον αφορά την υλοποίηση του συντονισμού, Ακούσαμε μια πολύ καλή ερώτηση για τη χρήση ψηφιακών λύσεων και για την ανταλλαγή δεδομένων. Πράγματι, έχουμε ένα σύστημα ανταλλαγής δεδομένων. Θα υπάρξει ένα εργαστήριο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Εκεί θα συζητηθεί η ανταλλαγή των δεδομένων και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες βιώσιμες λύσεις που να χρησιμοποιούνται ευρύτερα διότι όλοι μας θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο ελαχιστοποιεί τα ασφάλματα και αποκλείει τις ε, απάτες. Τώρα, όσον αφορά ε, το ελάχιστο ημερομίσιο, την ελάχιστη αμοιβή, δεν το ανέφερα αυτό το θέμα στην παρέμβασή μου. Όταν αναφερόμουν σε ίσες ευκαιρίες, εννοούσα ίσες ευκαιρίες, ίση πρόσβαση σε κεκτημένα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης. Όταν διέρχονται τα σύνορα οι άνθρωποι ούτως ώστε να μπορεί ο λαός να ωφελείται από τα κεκτημένα του δικαιώματα, ο Είναι λυπηρό πως ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό. Και το όλο θέμα της κοινωνικής κάλυψης και ένταξης εντάσσεται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα κοινωνικά ζητήματα θεωρώ ότι έχουν συζητηθεί εκτενώς πρόσφατα και τα κράτη-μέλη έχουν συμμετάσχει πολύ στις συζητήσεις. Είναι ευπρόσδεκτη αυτή η εξέλιξη και με χαροποιεί το ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και οι συστάσεις λαμβάνουν υπόψη ε, τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων κρατών μελών, ούτω ώστε οι συστάσεις να είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν και να ακολουθηθούν. Ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα σε ένα ελάχιστο εισόδημα εντάσσεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εντάσσονται αυτά τα ζητήματα. Επικρατούν διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν κάποια προγράμματα, κάποια πλαίσια για την ε, ελάχιστη αυτή αμοιβή με ένα εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα. Πιστεύω ότι για την ώρα αυτά είναι όλα όσα θα μπορούσα να σας πω. Είναι μια αρχική απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις σας και βέβαια αν έχετε και άλλες ερωτήσεις με τα χαράς να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Πρώτα απ' όλα για την άδεια μητρότητας και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι πολύ φιλόδοξη η πρόταση, την καλωσορίζουμε και θα ξεκινήσουμε την συγκεκριμένη συζητήσεις ε, κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, ε, αλλά όπως έχουν τώρα τα πράγματα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Αλλά βεβαίως θα συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο για να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις στο συντομότερο δυνατόν. Δεύτερον, υπήρξε μια ερώτηση από την κυρία Γιουγκέριους για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Βεβαίως είναι υψηλή πολιτική προτεραιότητα Γι' αυτό θέλουμε να το προωθήσουμε κατά την διάρκεια της Προεδρίας μας σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και βεβαίως το θέμα της χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικό και έχει τέθει πολλές φορές αλλά δεν είναι δική μου αρμοδιότητα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Νεολαίας Τώρα, για την απόσπαση εργαζομένων. Βεβαίως είναι ένα περίπλοκο και διχαστικό θέμα. από την άλλη, βεβαίως κάποιους ενώνει. Και λογικό είναι ότι τα κράτη-μέλη είναι υπέρ και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα και με τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείε μας. Και κατανοητό είναι ότι η, εταιρεία, η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς απαιτεί και την ορθή παροχή των υπηρεσιών και η ισορροπία που πρέπει να βρεθεί βεβαίως έχει συζητηθεί και εδώ και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εκμεταλλευτούμε και τα επιτεύγματα της προηγούμενης Προεδρίας και να βρούμε έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό. Απαιτείται να βρεθεί ένας συμβιβασμός ε, και απαιτείται συμβιβασμός από όλες τις πλευρές, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος η οδηγία αυτή να μην εφαρμοστεί πριν από το τέλος της ε, εντολής ε, της θητείας του Κοινοβουλίου το 2019. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε το θέμα και στο Συμβουλίο του Οκτωβρίου. Είναι λοιπόν υψηλή προτεραιότητα για μας και δεν ξέρω αν θα ικανοποιηθεί κανένας πλήρως με το αποτέλεσμα. Έτσι είναι οι συμβιβασμοί, αλλά πρέπει να πετύχουμε έναν συμβιβασμό. Και έρχομαι έτσι στα γενικότερα θέματα που έθεσε ο κύριος Κάσα και άλλοι για την γενική ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώ αναφέρθηκε η διαφορά μεταξύ παλιών και νέων κρατών μελών και όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό τώρα να έχουμε πολιτική ενότητα παρά ενότητα σε κάποιες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες. Νομίζω λοιπόν ότι μια φορά ως επιλογή μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού συμφέροντος. Η πραγματική επιλογή είναι μεταξύ εθνικού και κοινού συμφέροντος και των Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το ευρωπαϊκό συμφέρον ως κοινό συμφέρον και άρα και ως εθνικό συμφέρον. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγκρούεται το βραχυπρόθεσμο με το μακροπρόθεσμο συμφέρον των κρατών μελών. Και αν δούμε τους δύσκολου καιρού της Ευρώπης στο παρελθόν, ε, ε, εδώ και 10 χρόνια πηγαίνουμε από τη μία κρίση στην άλλη, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πίεση μεγάλη για τα βραχυπρόθεσμα και τα θέματα που είναι στενού εθνικού συμφέροντος, αλλά νομίζω ότι ε, περνάμε σε μια πιο αισιοδοξή εποχή και υπάρχει μια δυνατότητα ακριβώς να ξεκινήσουμε να προωθούμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πιο γρήγορα και με πιο ενωμένο τρόπο. Μπορούμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την συγκυρία και να αρχίσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο αμέσω. Κάποιοι έχουν ζητήσει τον λόγο. Τόμας Μαν πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας στηρίζω ειδικά όταν λέτε ότι έχουμε μεγάλες ελπίδες από την Εστονία. Είχαμε πλήρη την αίθουσα της Ολομέλειας ε, στο Στρασβούργο γιατί έχουμε μεγάλες προσδοκίες από εσά γιατί είστε δυναμική χώρα και έχετε την σωστή προσέγγιση. Είπατε πως υπάρχουν ε, μεγάλες δυσκολίες στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε μια ευκαιρία μπροστά μας. Θεωρώ το βραβείο Καρλομάγνου θα έπρεπε να χωριστεί σε δύο μέρη και να τιμήσουμε τον κύριο Τραμπ και την κυρία Μέη γιατί όσο υπάρχει απειλή του προστατευτισμού και της σκληρής γραμμής της κυρίας η οποία κυβερνά στη Μεγάλη Βρετανία ξεκαθαρίζει το ότι οι υπόλοιποι 27 πρέπει να συνεργαστούμε. Λοιπόν, και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους Βρετανούς συναδέλφους οι οποίοι προσεχώς θα απουσιάζουν από αυτή την υπόθεση. Επίσης, όταν λέτε περισσότερη Ευρώπη και όχι περισσότερο να επικεντρωνόμαστε στα κράτη-μέλη. Για την ψηφιακή Ευρώπη δεν αρκεί να λέμε ότι θα συνεχίσουμε. Επίσης, για το μέλλον της εργασίας. Κάποιοι από εμά είχαν πάει στην Silicon Valley για να δούμε από κοντά το πώς θα έχει η δουλειά, η εργασία του μέλλοντος. Ε, θα θέλαμε λοιπόν συγκεκριμένες ε, προτάσεις και παραδείγματα. Και το επόμενο, ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, υφίσταται επίθεση. Οι μεν λένε ότι είναι λόγια χωρίς αντίκρισμα και οι δε λένε ότι είναι βαθιά παρέμβαση στα δικαιώματα των κρατών μελών. Λοιπόν, μια ισορροπία νομίζω θα ήταν να πούμε πάρτε το σοβαρά, κάντε μια εντατική συζήτηση, φροντίστε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για να μην αποκοπεί ο κόσμος από τις μεγάλες κοινωνικές ε, διεργασίες. Πρόκειται λοιπόν για μια καλή ιδέα και θα πρέπει ε, να σταματήσουμε κάποτε να μιλάμε για αυτό το διχασμό Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Ε, να οικοδομήσουμε γέφυρες. Νομίζω αυτή ήταν η σωστή θέση ε, βασιζόμαστε λοιπόν ε, σε εσά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελίζαμπεθ Μονάνσοτιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία και κύριε Υπουργέ, καταρχάς κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Έχουμε πολλές ε, μεγάλες προσδοκίες από την Προεδρία σας. Ιδιαίτερα για το θέμα το οποίο, με για το οποίο είμαι υπεύθυνοι μαζί με όλους τους κοιόδης εισηγητές, γιατί κάθε πολιτική ομάδα έχει πολύ σημαντική, σημαντικό ρόλο για να δημιουργηθεί αυτή η ενότητα στην οποία αναφερθήκατε και για να υπερβούμε τους ε, διχασμούς, γιατί ο διχασμός είναι κάτι που πρέπει να ανήκει στο παρελθόν. Το μέλλον πρέπει να είναι η σύγκληση και η συνοχή μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αναφερθήκατε λοιπόν στην ενότητα. Αυτή είναι επιδιώκουμε εδώ ως Κοινοβούλιο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την επιτύχουμε μέσω πνεύματος συμβιβασμού. Αλλά υπάρχει το Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο, για το οποίο είστε υπεύθυνοι τώρα, για μερικούς μήνες. Στο Συμβούλιο λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω, να σας οικετεύσω ε, να προσέξετε τα εξής. Το πρώτο είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. τον Ιούνιο παραλίγο να επιτευχθεί συμφωνία υπό την Μαλτέζικη Προεδρία στο Συμβούλιο. Σήμερα θα μπορούσατε να δεσμευτείτε ενώπιόν μας να καταλήξουν με συμφωνία οι συζητήσεις στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Γιατί οποιαδήποτε κόλληση εργία στο Συμβούλιο είναι πολύ κακός για την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Δεύτερον, η συνάδελφος ε, Αγνές Γιονγκέρους που είναι συνεισηγήτρια το ανέφερε είπε ότι θα ξεκινήσετε πρέπει να ξεκινήσετε τον τριμερή διάλογο. Εγώ είμαι ακόμη πιο απαιτητική. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου υπό την Προεδρία σας. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό μπορεί να ξαναδώσει ελπίδα στο σύνολο των Ευρωπαίων συμπολιτών μας για μια Ευρώπη που σήμερα πρέπει να γίνει πραγματικά κοινωνική Ευρώπη. Γιατί και με το κείμενο αυτό και με τα άλλα που ανέφεραν οι συνάδελφοί μου, δημιουργούμε μια βάση της κοινωνικής Ευρώπης. Βεβαίως, ε, η νομική βάση του 1996 αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Αλλά τι περιμένουν σήμερα όλοι οι συμπολίτες μας. Θέλουν το πρόβλημα της απασχόλησης να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η προώθηση της κοινωνικής Ευρώπης παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Θέλω λοιπόν και στο χρονοδιάγραμμα και στην επιτυχία των τριμερών διαλόγων και στο πνεύμα, στην προώθηση του πνεύματος της κοινωνικής Ευρώπης, σε αυτά τα θέματα έχουμε πλήρη επιτυχία στην Προεδρία σας, κυρία και κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος Ενρίκε Καλβέ Τσαμπών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και σίγουρα δεν είναι η τελευταία φορά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Θέλω να είμαι απόλυτα συγκεκριμένος. Όλοι συμφωνούν, δεν επιμένω, ότι τώρα έχει γίνει σαφές ότι για να έχουμε την κρίσιμη μάζα που χρειαζόμαστε, την κρίσιμη μάζα στήριξης μεταξύ των συμπολιτών μας, πρέπει να στραφούμε πολύ περισσότερο προς τα κοινωνικά θέματα και πλησιάζουν και οι εκλογές. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να θεωρούμε θα απορισμένους ως μια οικονομική ελίτ χαμένη κάπου. Πρέπει να υπάρξει μια στροφή προς τα κοινωνικά θέματα, όλοι συμφωνούμε. Λοιπόν, αυτό το είναι γνωστό. Αλλά αυτό όμως δεν πρέπει απλώς να μεταφραστεί σε γενικόλογες διακηρύξεις περί ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και άλλες ε, καινολογίες. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχει η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με ένα σχέδιο, μια αντίληψη για κοινωνικές δράσεις που θα πρέπει να βασίζονται στις αξίες μας. Το βασικό είναι να επιτύχουμε 2, 3, 4 συγκεκριμένα αποτελέσματα που να αφορούν τους περισσότερους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι η Κομισιόν έκανε λάθος ξεκινώντας με ένα θέμα που τελικά μας διχάζει περισσότερο. Ενώ δεν είχαμε ακόμη αποτιμήσει την προηγούμενη εκδοχή, την εφάρμοσαν εν πάση περιπτώσει οφείλεται σε εκλογικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα τώρα αυτό έχει περάσει. Οπότε, είστε διατεθειμένοι να απαιτήσετε στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν να δημιουργηθεί ένα είδος προγράμματος δράσης ρεαλιστικό και εφικτό, όχι να τα θέσετε όλα μαζί σε θέματα που πραγματικά αφορούν όλους, όπως για παράδειγμα το ελάχιστο εισόδημα ένταξης όπως το, όπως λέμε. Όπως για παράδειγμα η δημιουργία καλών θέσεων εργασίας και η καλύτερη χρήση του εύση γιατί η απασχόληση είναι ο πρώτος λόγος για την ανισότητα. Πώς θα πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα για να καταπολεμήσουμε όλες τις ανισότητες μέσω μέτρων αλληλεγγύης για να, για να καταπολεμήσουμε την ένδυα πρέπει να θέσουμε ορισμένες προτεραιότητες για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα πριν το 2019, κάτι που να γίνει αντιληπτό. Βεβαίως να έχουμε καλές προθέσεις και να προωθήσουμε ε, μεγάλα προγράμματα, να αποφύγουμε τα δευτερεύοντα που μας ε, χωρίζουν. Πέρα από τις ε, διοργανικές ε, διακηρύξεις που θα είναι πολύ ευχάριστες, αλλά μόνο ευχάριστες, το βασικό είναι να πούμε Μέχρι το 19 θα κάνουμε αυτό. Καταπολέμηση τη ε, φτώχεια με τα εξή μέτρα. Το ελάχιστο εισόδημα που θα μπορέσει να αξιοποιήσει η Προεδρία για να διευκρινίσουμε ότι το ελάχιστο εισόδημα δεν είναι να κάνει με τις ελάχιστες απολαβές. Αυτό να είναι σαφές. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα αποτελεσματικά ζητήματα. Μπορεί να εστιάσει εκεί η Προεδρία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία και τον κύριο Υπουργό για τις ε, πληροφορίες. Είναι σαφές ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η Προεδρία σας και σίγουρα έρχεται σε μια στιγμή που σίγουρα θα δημιουργήσει έντονο φόρτο εργασίας. Αλλά είναι πολύ ουσιώδης η συγκυρία για τα θέματα που μας απασχολούν εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη είναι μέσα σε μια περίοδο δύσκολη οικονομική και πολιτική λόγω του Brexit. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι πώς αντιλαμβάνονται την Ένωση οι συμπολίτες μας και ένα μη αμεληταίο τμήμα των συμπολιτών μας απομακρύνεται από το ευρωπαϊκό εγχείρημα γιατί θεωρεί ότι το εγχείρημα αυτό είναι πολύ απομακρυσμένο από την καθημερινότητά τους. Όταν ρωτάμε τους πολίτες ε, τι τους ανησυχεί είναι η απασχόληση, αλλά και η ποιότητα της ε, απασχόλησης και η κοινωνική ασφάλιση. Αυτά είναι τα θέματα. Και η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες μορφές εργασίας τους ανησυχεί. Εδώ έχει ανοίξει λοιπόν ένα παράθυρο ευκαιρίας. Μία δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα, ε, μία ελάχιστη βάση κοινωνικών δικαιωμάτων. Αλλά αυτό το παράθυρο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αν δεν το αξιοποιήσουμε θα είναι απλώς ένα ανοιχτό παράθυρο από όπου θα δημιουργηθεί ρεύμα αέρα που θα κάνει τους ανθρώπους να κρυώσουν προς την Ευρώπη. Σας καλώ λοιπόν και ελπίζω πραγματικά να βασιστείτε στους κεντρικούς πρωταγωνιστές που είναι η κοινωνική εταίροι, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και των μισθωτών. Αυτή θα είναι η βάση αυτού του τόσο δύσκολου αλλά αναγκαίου συμβιβασμού για τα διάφορα θέματα που μπορούν όντως να μας οδηγήσουν σε ε, συμβασμούς που δεν θα είναι ο ελάχιστος κοινό παρνομαστής, αλλά με πολύ περιεχόμενο. Ευχαριστώ για να τόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαν να παίρνω τηλέφωνο τώρα στο ραδιόφωνο και να ζητάω να ευχηθείτε χρόνια πολλά στον άντρα μου που είναι στην κουζίνα και θα ευχαριστηθεί που θα τα ακούσει. Ξέρετε, σε κάθε προεδρία λέμε ότι ελπίζουμε ότι η Προεδρία σας θα επιτύχει τρομερά πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο εξάμεινο. Ως Επιτροπή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και η επικουρικότητα. Ορισμένες φορές με τη συνάδελφο Ενρίκη και καπνίζουμε στο καπνιστήριο και συζητάμε τι είναι η επικουρικότητα. Οπότε να σας κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι τα λιγότερο επίμαχα θέματα που θέλετε να προωθήσετε για να μην κολλήσουμε σε αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό σίγουρα δεν είναι το ελάχιστο εισόδημα. Ίσως κάτι που να έχει να κάνει με την μπλε κάρτα, με την αδήλωτη εργασία. Πού θεωρείτε ότι υπάρχει κοινή καλή θέληση μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή, για ποια θέματα θεωρείτε ότι δεν θα σκοτωθείτε στο Συμβούλιο. Με συγχωρείτε που τα λέω έτσι αδρά. Και κάτι άλλο που είπε η Μαρτίνα και με το οποίο συμφωνώ. Ναι, βεβαίως. Η Εστονία έχει επιτύχει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές συνταγέ, ε, οι ρυθμίσεις για την ε, γονική άδεια, όλα αυτά είναι θαυμάσια. Και θα αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία για να κάνετε γνωστά τα επιτεύγματά σα και σα εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχω δύο διαφορετικά θέματα που θα, θα αναθέσω. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε στην μπλε κάρτα που αφορά τα δικαιώματα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρώπων με πολλές δεξιότητες, Ε, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών είναι αρμόδιο γι' αυτό. Από πλευράς απασχόλησης, πώς μπορεί να συμμετάσχουν οι ασχολούμενοι την απασχόληση σε αυτή τη συζήτηση και στους τριμερείς διαλόγους που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν αρκετά σύντομα. Διότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ότι σχετίζεται με μετανάστευση εργαζομένων να αντιμετωπίζεται σαν θέμα φραγμών και όρους εισόδου παρά τι ωφέλη αποκομίζει αυτό για την αγορά εργασίας και πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Εσείς, α, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε πλευράς ε, φορέων που ασχολούνται με την εργασία σε αυτό το θέμα. Μετά, που πρέπει να ηγηθούμε. Έχουμε δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουμε να ηγηθούμε στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η Προεδρία σας, πώς θα κινηθεί σε αυτόν τον τομέα. Στα πλαίσια της απασχόλησης, ε, πώς θα οδηγηθούμε σε αυτή τη μετάβαση που συζητούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον ΟΗΕ και το αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας. Πώς μπορείτε να προωθήσετε τη διά, διάσταση της απασχόλησης προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε κάποιες ε, δεξιότητες και αν δεν προσελκύσουμε τους ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες δεν θα καταπολεμήσουμε το κλίμα και δεν θα ηγηθούμε στον τομέα και δεν θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και το εργατικό δυναμικό δεν θα συμμετάσχει με τον κατάλληλο τρόπο στι αναγκαίε αλλαγέ. Ευχαριστώ. Θέλω και το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν άλλον όμω. Οπότε κλείνουμε τις ερωτήσεις και παρακαλώ τους δύο υπουργού ποιος θέλει να πάρει το λόγο πρώτος ή κυρία Υπουργό, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, διότι εκφράσατε την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ επίσης και για τις ερωτήσεις. Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως ότι δεν είναι εύκολη η καιρή αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρουσιάζονται και κάποιες ευκαιρίες. Ευκαιρίες για να γίνει αντιληπτή η αξία της ενότητας. Και ίσως αυτό θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους να προσπαθήσουν να πετύχουν κάτι. Η Προεδρία μας με τις πρωτοβουλίες της όπως είναι ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων ε, έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι καινούριο, κάτι σημαντικό. Όσον αφορά την ενότητα της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικά τα κοινωνικά ζητήματα διότι τα κοινωνικά θέματα είναι εύληπτα για τον κόσμο. Όσο καλύτερα αντιμετωπίζονται τα κοινωνικά ζητήματα στα κράτη-μέλη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπιστοσύνη του λαού προς την κυβέρνηση και προς την Ευρώπη. Και είναι καθήκον μας να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά τα θετικά παραδείγματα του τι μπορεί να επιτευχθεί σε μια περίοδο που υπάρχουν διαφορές μεγάλες μεταξύ κρατών μελών, σωστά το λέτε. Ε, δεν είναι εύκολο να βρούμε τα σωστά μέτρα σε αυτό το τομέα πολιτικής. Ίσως μέσω του κανονισμού συντονισμού μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες ευκαιρίες. Τα ατομικά δικαιώματα για ανθρώπους με μικρά παιδιά. Εκεί υπάρχει περιθώριο συμφωνίας. Αυτό που θα ήθελα να κάνω κατά τη διάρκεια της Προεδρίας είναι μια σοβαρή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Να εξετάσουμε πρακτικές λεπτομέρειες να δείξουμε κάποια αποτελέσματα που θα ενθαρρύνουν ε, ε, νέο προβληματισμό, νέα προσέγγιση στα κράτη-μέλη. Σαν ένα τμήμα του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε διαβούλευση για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι καρποί αυτής της διαβούλευσης. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών ε, δικαιωμάτων καλύπτει, περιλαμβάνει το δικαίωμα σε ένα ελάχιστο εισόδημα. Οπότε αναπόφευκτα θα το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αυτά έχω να πω και θα δώσω το λόγο τώρα στον συναδελφό μου. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το θέμα της απόσπασης ε, των εργαζομένων και το χρονοδιάγραμμα. Θέλουμε μέχρι τον Οκτώβριο να καταλήξουμε σε γενική προσέγγιση και αν είστε έτοιμοι ξεκινάμε αμέσως στον τριμερή διάλογο και οι δυνατόν δεν θα είχαμε πρόβλημα να ολοκληρωθούν επί προεδρίας μας οι τριμερείς διάλογοι. Το πρώτο βήμα είναι να έχουμε έτοιμο στο Συμβούλιο, να έχουμε έτοιμη τη γενική προσέγγιση τον Οκτώβριο. Τώρα η μπλε κάρτα Παρακολουθούμε τις εξελίξεις εκ του σύνεγγης στο Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, αλλά δεν σχεδιάζεται κάποια συζήτηση σε επίπεδο το, του Συμβουλίου Υπουργών Εργασίας. Τώρα, σχετικά αφορά ε, τις μελλοντικές εργασίες, αυτές αναφέρθηκαν σε πολλές ερωτήσεις, όπως σας είπα. Τώρα, το πώς θα γεφυρώσουμε την μεταμόρφωση της κοινωνίας και την καινοτομία και πώς θα ενταχθούν όλα αυτά στα κοινωνικά συστήματα, αυτές οι αλλαγές είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Η πράσινη οικονομία, ε, η αλλαγή αυτής ή η ψηφιακή οικονομία. Ε, και εδώ βλέπουμε καμιά φορά λόγω της μειώσης της κοινωνικής προστασίας ότι υπάρχει η δυσκολία της μετάβασης για τους εργαζομένους. Υπάρχει και το πρόβλημα της περιφερειακής πολιτικής, διότι κάποιες περιφέρειες των παλαιών οικονομιών δεν θα είναι ίσως ε, ε περιφέρειες της νέας οικονομίας. Δεν είναι αυτός ένας λόγος για να σταματήσει η πρόοδος, είναι ένα πρόβλημα προς επίλυση. Και στον εκεί Προεδρία θα κινηθεί και στα δύο πεδία. Θα εστιαστούμε στην ψηφιακή καινοτομία, θα προωθήσουμε αυτόν τον τομέα, ταυτόχρονα όμως θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να μετασχηματίσουμε την κοινωνική μας πολιτική, ούτως ώστε να είναι επαρκής για τις νέες ανάγκες που απορρέουν από τη νέα ε, ψηφιακή κοινωνία. Αυτό πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό εστιαζόμεθα ως Προεδρία επί της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και της ελεύθερης διακίνησης δεδομένων για κάθε Ευρωπαίο πολίτη, που θα μπορεί να ωφελείται τις νέες τεχνολογίες ο πολίτης. Ταυτόχρονα είναι σημαντικότατο να εξετάσουμε το τι πρέπει να γίνει από την κοινωνική πλευρά για να προστατεύσουμε επαρκώς ε, τους πολίτες για να γίνει με επιτυχία μετάβαση. Ίσως αυτό μπορεί να δώσει μια νέα ορμή στην προσπάθεια για ενότητα. Αυτή ε, η πρόταση για τον κοινωνικό πυλώνα. Σε τεχνικό επίπεδο μπορούν να συζητήσουν κάποιοι αν αυτό είναι αρκετά φιλόδοξο ή αν η διατύπωση της αρχής είναι η βέλτιστη δυνατή. Αλλά είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει τις βασικές αρχές ή να θεωρήσει ότι δεν είναι κοινέ αρχές ε, για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Αναφέρονται σαφώς όλα αυτά και χρειάζεται πολιτική δέσμευση να προωθηθεί αυτός ο πυλώνας που είναι ενωτική βάση για τις μελλοντικέ ε, συζητήσεις. Αυτά και σας ευχαριστώ. Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τη συζήτηση. Θεωρώ πως η εισαγωγή στην Προεδρία σας ήταν μια καλή αρχή. Τότε βλέπω η Προεδρία σας ε, έχει αναλάβει πολλά πράγματα και στον δικό μας τον τομέα και ελπίζω να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που θα προωθήσουν την Ευρώπη στα θέματα μας. Δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερος ε, που θα ενισχύσουν την Ευρώπη. Το θέμα ε, το ένα είναι ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Κανείς δεν ξέρει τι συγκεκριμένες επιπτώσεις ή αποτελέσματα θα έχει αυτή η διακήρυξη. Ελπίζω να στηρίξετε την θέση της Επιτροπή μας πως ε, θα είναι κάτι παραπάνω από ε, μεγάλα λόγια και πανηγυρική αλλά θα βοηθήσει να γίνει η Ευρώπη πιο κοινωνική και βεβαίω συχνά υπάρχει μια παρεξήγηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα δεν είναι να στηρίξουμε τις χώρες που έχουν ασθενέστερο κοινωνικό κράτος και επίπεδο για να έρθουν στο επίπεδο των άλλων χωρών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για να είναι απτή η κοινωνική Ευρώπη σε ολόκληρη την Ευρώπη σε μια διαδικασία σύγκλησης που θα ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Η δεύτερη παρατήρηση. Βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση για το θέμα της απόσπασης. Σε δύσκολη θέση. Και εδώ υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις. Το συζητήσαμε και στο Συμβούλιο. Η αρχή ίση αμοιβή για ίση εργασία δεν σημαίνει να ε, υπάρξει μια εξίσωση μισθών στην Ευρώπη. Εγώ ως συνδικαλιστής ε, και ο Κλοντρολέν και, και ο Γκέρις οπωσδήποτε θα με στήριξουν για να δούμε ακριβώς το πώς ε, θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια άνοδο των μισθών σε εθνικό επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ αντίσταση σε αυτό το θέμα. Και όταν μιλάμε για ένα ελάχιστο εισόδημα, οπωσδήποτε εγώ θα χαιρόμουν εάν ε, συζητούσε η Εστονική Προεδρία όχι έναν ενιαίο βασικό ευρωπαϊκό μισθό στην Ευρώπη. Δεν στέκει αυτό αλλά έναν ε, βασικό μισθό ανά χώρα που θα ταιριάζει στο επίπεδο της χώρας για να μην είναι ο κόσμος φτωχός. Αυτό νομίζω θα μπορούσε να προκύψει από την συζήτηση για να ενισχυθούν τα κοινωνικά δικαιώματα και χωρίς ιδεολογίες, απλά ανατολισμένοι, προς το συμφέρον των ανθρώπων και ειδικά των φτωχότερων στην Ευρώπη που είναι αρκετοί. Εάν λοιπόν ε, πάει προς αυτή την κατεύθυνση η συζήτηση στην Προεδρία σας, εγώ θα χαιρόμουν. Οπωσδήποτε μπορώ να σας υποσχεθώ την καλή συνεργασία της Επιτροπής μας. Έχουμε πολλά να κάνουμε στην Ευρώπη. Πριν ε, βυθιστεί λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. So, dann haben wir etwas... Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο τώρα πριν συνεχίσουμε. Θα παραδώσω τώρα την Προεδρία στη Μαρίτα. Σας χαιρετώ. Καλές διακοπές, εύχομαι. Αλήξη και ξεκούραση. Και υγεία. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους συνεργάτες εδώ. Okay, friends. Καλώς, φίλοι μου. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καταρχάς, ορίζω εκείνους από εσά που είστε ακόμα εδώ και αυτούς που δεν είναι εδώ. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ παρά το γεγονός ότι είναι η τελευταία ημέρα πριν τις διακοπές μας, τις διακοπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή η ακρόαση αφορά τη δεύτερη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα καρκινογόνα και τα μεταλλαξιογόνα και τη σχετική οδηγία. Ήταν καρποφόρο το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου και πάμε στο δεύτερο γύρο. Αυτή η πρόταση ακολουθεί την πρώτη και ίσως να είναι κάπως ε, δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς λεπτομέρειες, διότι έχουμε δύο χαρτοφυλάκια για την ίδια οδηγία, ε, παράλληλες πορείες με κάποια άλλη επικάλυψη, θα τα καταφέρουμε. Ήταν σαφής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φιλοδοξία είναι να γίνουν και πολλές αναθεωρήσεις του παρατήματος 3 της οδηγίας για τα καρκινογόνα και τα μεταλλαξιογόνα, διότι υπάρχουν περισσότερες ουσίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και το περιμένουμε αυτό. Έχουμε σήμερα μιλητές από το ETUC, από το SCOWEL και από την Business Europe. Θα μας μιλήσουν ε, για το θέμα, θα εκφράσουν τις απόψεις τους, θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις μας και σας ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να έρθετε και χαιρόμαστε που ο Επίτροπος Τάισεν είναι εδώ μαζί μας για να παρουσιάσει η Επίτροπος τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα ακρηγορήσω Βέβαια είναι σημαντικό για μας να έχουμε τον αρμόδιο υπουργό παρόντα που εκπροσωπεί την Προεδρία, τον κύριο Οσινόφσκι, που είναι εδώ από την αρχή, στην αρχή των συζητήσεων πρέπει να αποχωρήσει αργότερα όμως και ελπίζουμε ότι αυτή η εισαγωγή να βοηθήσει και την Προεδρία να κινηθεί γρήγορα και να λάβει σωστές αποφάσεις. Επίσης θέλω να κλείσω ευχαριστώντας όλους για το επιτελεστέν έργο κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συζητήσεων για την οδηγία. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό και αυτό πρέπει να πω ότι μας δίνει ε, περισσότερο θάρρος και κουράγιο να πολεμήσουμε. Ε, έχουμε τα γνωστά πρόσωπα από την Επιτροπή Απασχόλησης. Προσβλέπουμε τα επόμενα θέματα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Τάισον. Παρακαλώ να μας κάνετε μια εισαγωγή για τα θέματα που θα συζητήσουμε σε αυτό το δεύτερο γύρο. Καλώς, ευχαριστώ, λέει η κυρία Τάισαν, αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Και αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κύριο Σινόφσκι, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη και ξέρετε ότι στην ακρόασή μου ήδη προσωπικά δεσμεύτηκα να καταπολεμήσω τον ε, καρκίνο που προξενείται από, στο χώρο εργασίας. Ε, προσπάθησα να επικαιροποιηθεί η οδηγία για τα καρκινογόνα και τα μεταλλαξιογόνα που είχε αποτελματωθεί, ετελούσε πνώση επί σειρά ετών Χαίρομαι που στη πρώτη φάση ε, συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για ε, τις αναγκαίες αλλαγές και το συζητήσουμε τις επόμενες. Σας συγχαίρω, κυρία Πρόεδρε, ήσασταν εισηγήτρια για, την, ε, για τα πρώτα μέτρα. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τα επιτευθέντα αποτελέσματα και η Εσθονική Προεδρία θέλει να προωθήσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Σήμερα ξεκινούν οι συζητήσεις για τη δεύτερη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μαζί με την πρώτη θα βοηθήσει να σωθούν ζωέ πάνω από 100.000 ε, εργαζομένων για τα επόμενα χρόνια. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής οδηγίας, ε, καλύπτει ε, και διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μηχανές εσωτερικής καύσεως και τα αλάδια Λοιπόν, οι μηχανικοί που αλλάζουν τα λάδια σε μηχανήματα, ε, σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα θα μπορούσαν να ε, γλιτώσουν από τον καρκίνο του δέρματος λόγω της προτάσεως. Έχουμε και νέα όρια επαγγελματικής έκθεσης για πέντε καρκινογόνες ουσίες, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα για ε, τις διάφορες ουσίες. Έτσι θα αλλάξει η προστασία, τα μέτρα προστασίας που ισχύουν στα κράτη-μέλη και για κάθε ένα από τα καρκινογόνα περίπου 20 κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν χαμηλότερα εθνικά όρια, εθνικές οριακές τιμές. Μέλη του Κοινοβουλίου πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στην καταπολέμηση του καρκίνου του δημιουργείται στον επαγγελματικό χώρο και χρειαζόμαστε νομοθεσία που θα κάνει τη διαφορά και που θα είναι αποτελεσματική επιτόπου Καταρχάς αυτό σημαίνει ότι σε αυτόν τον πολύ τεχνικό τομέα η σωστή προστασία των εργαζομένων μπορεί να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά μόνο να ακούσουμε τους επιστήμονες που κατανοούν καλύτερα πώς οι καρκινογόνες ουσίες επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων. Δεύτερο αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και συμβουλές από τους κοινωνικούς εταίρους. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών γνωρίζουν καλύτερα το πώς χρησιμοποιούνται αυτέ οι επικίνδυνε ουσίε στον χώρο εργασία και ποια προστατευτικά μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Ξέρετε ότι η υλοποίηση των προτάσεών μα είναι κάτι που θέλουμε να προωθήσουμε διακαώ. Δεν ε, έχει νόημα να ετοιμάζουμε μέτρα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Άρα έρχομαι στο παράδειγμα των καυσίμων δίζελ. Κάποιοι που σας θα περιμένετε να τα δείτε σε αυτή τη δεύτερη πρόταση να καλύπτονται. Προσεκτικά το εξετάσαμε το θέμα αλλά έπρεπε να συμπεράνουμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή, και λέω αυτή τη χρονική στιγμή, η θέσπιση μέτρων για τα καύσιμα ντίζελ δεν θα ήταν κάτι αποτελεσματικό, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα καθορίσουμε την ουσία με τέτοιο τρόπο που να είναι προσμετρήσιμη στον τόπο εργασίας. Περαιτέρω μελέτες χρειάζονται για το diesel, αλλά αυτό βεβαίως δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις προσπάθειες σε ουσίες όπου υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Βασίζουμε στην στήριξή σας να προωθήσουμε γρήγορα αυτή τη δεύτερη ε, πρόταση με την ομάδα μέτρων. Σας διαβεβαιώνω μέλη του Κοινοβουλίου ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα σταματήσει εδώ στη δεύτερη πρόταση. Ξεκινήσαμε προπαρασκευαστικές εργασίες για τη νέα ομάδα ουσιών και θα υποβάλουμε σχετική πρόταση για αυτές αρχές του επομένου έτους, αρχές του 2018. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αξιολογήσει και την ανάγκη να συμπεριλάβουμε και αναπαραγωγικές ουσίες ε, σε αυτόν τον τομέα. Το Κοινοβούλιο έχει ε, εκφράσει ανησυχή σε αυτόν τομέα και για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες ισχύει αυτό και θα πρέπει να καταλήξουμε σε στρατηγική, να αξιολογήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται από αυτές τις ουσίες και να βρούμε το καλύτερο μέσο για να εξασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των εργαζομένων της Ευρώπης και την προστασία των πολιτών. Ο καρκίνος σχετίζεται με την εργασία, είναι πραγματική τραγωδία για τους εργαζόμενους και για τις οικογένειές τους και ταυτόχρονα είναι και μεγάλο άχθος για όλη την κοινωνία. Μαζί μπορούμε να κάνουμε σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της ασθενείας. Βασίζομαι πάνω σας να σημειώσουμε καλή πρόοδο και σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, ώστε σύντομα να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις και στον κρότορο λαό τον εισηγητή και στους και εισηγητές και σε όλους σας εύχομαι ε, κάθε επιτυχία σε αυτή σας την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Τάισεν και τώρα θα δώσω το λόγο στον Υπουργό της Εστονίας που είναι επιφορτισμένος, είναι αρμόδιος για τα θέματα. Ο κύριος Σινόφσκι. Κύριο Σινόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χτες μόλις ε, το Συμβούλιο έκανε τις ε, προσωρινές ε, συμφωνίες για τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Νομίζω πως αξίζουν συγχαρητήρια. Βεβαίως δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Όπως ξέρετε η συμφωνία για το πρώτο μέρος ήταν συμβιβασμός με κάθε έννοια της λέξης. Όλοι έκαναν συμβασμούς. Και βεβαίως αυτό ήταν αναγκαίο για να προχωρήσουμε. Δεύτερον, δεν είναι τώρα η στιγμή για να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας. Όπως είπε και η Επίτροπος, η Κομισιόν εξετάζει το τρίτο πακέτο καρκινογόνων ουσιών με την τριμερή συμβουλευτική επιτροπή και το θέμα αυτό βέβαια είναι ψηλά στην ατζέντα Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εγώ θα σας παρακαλούσα να συνεχίσετε να το έχετε αυτό ως πρώτη προτεραιότητα, όπως φάνηκε και η σημερινή ακρόαση η εμπειρία βεβαίως ε, του πάνελ ε, δείχνει πως θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σε ευχαριστήσω όλους που αποδίδετε την σημασία που αξίζει στο θέμα αυτό και σας διαβεβαιώ πως από την πλευρά του Συμβουλίου είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει για το δεύτερο πακέτο όταν θα είστε έτοιμοι στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ε, τώρα ε, ε, να φύγετε βεβαίω, αλλά αναμένουμε την συνέχεια της προεδρίας σας και είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε κάποιους λόγους να επανέλθετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά έχουν τώρα την δυνατότητα οι βουλευτές να ζητήσουν το λόγο. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Καταρχάς θέλω να σας ακούσω, να ακούσω τις παρεμβάσεις, να ακούσω τους συναδέλφους και μετά κυρία Πρόεδρε θα λάβω το λόγο στο τέλος για να πω κάποια πράγματα για τις μελλοντικές μας εργασίες. the coordinators, Madam McIntyre, would you like to say something? Thank you, Madam President. Um, I think on behalf of the ECR, I would like to... Σας ευχαριστώ, κυρία Μακίντερ. Σας ευχαριστώ εξ όνομα του ECR. Θα μπορούσαμε να διευρύνουμε, θα έλεγα, το δεύτερο αυτό κείμενο της οδηγίας τα όρια που περιέχονται σε αυτές τις προτάσεις της ε, Κομισιόν βασίζονται σε δουλειά ετών της ε, Κομισιόν και πρέπει νομίζω να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια τάση για εμάς τους ε, έρασιτέχνες που εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των πολιτών να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία και να βασιζόμαστε σε αυτά στο μέτρο του δυνατού. Μέρος της επιτυχίας αυτών των οδηγιών, γιατί βεβαίως μιλάμε για πολλές οδηγίες, Ε, είναι το ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση, να μειώσουμε τον αριθμό των θανάτων και αρρωστιών από την έκθεση σε καρκινογόνα σε άλλε, και σε άλλες επικίνδυνες ουσίες. Το κλειδί εδώ λοιπόν είναι να φροντίσουμε να έχουμε κάποια όρια τα οποία θα είναι μετρήσιμα στο χώρο εργασίας. Μια φορά προτείνουμε πράγματα τα οποία είναι πέρα από το τι είναι δυνατόν. Και φοβάμαι ότι καμιά φορά θα χάσουμε τον σεβασμό των ανθρώπων που ξέρουν τι λένε με το να λαμβάνουμε αυθαίρετες αποφάσεις. Δεν λέω ότι έχουμε φτάσει εκεί, θεωρώ ότι καλά τα πάμε μέχρι στιγμής, αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ε, μιλάμε για έκθεση στον χώρο εργασίας σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες και πρέπει η έμφαση να είναι στην εφαρμογή ελέγχων στο χώρο εργασίας και ορθών πρακτικών για να προστατεύουμε τον κόσμο από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Τελικά λοιπόν θα πρέπει πάντα να επιδιώκουμε να επιτυχάνουμε το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Ε, χαμηλότερο ακόμα και από αυτό που ορίζει η νομοθεσία. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επενδύσουν σε έρευνα και να ενθαρρύνουμε βεβαίως ε, την προσπάθεια για συνεχώς χαμηλότερο επίπεδο, αλλά να μην καθορίζουμε αυθαίρετα όρια τα οποία θα είναι πολύ χαμηλά και άρα ανεφάρμοστα. Να ενθαρρύνουμε λοιπόν την ε, διαδικασία μείωσης της έκθεσης και να ενθαρρύνουμε τις εταιρείε να πάνε κάτω από το όριο που καθορίζει ο νόμος ε, είναι ε, κάτι το θετικό. Δηλαδή αυτό το όριο είναι αυτό το οποίο ορίζει ο νόμος, αλλά αν μπορούν να κάνουν και κάτι καλύτερο, βεβαίως. Και αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, θεωρώ πως η αναλογικότητα και το εφικτό του πράγματος πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οπότε οποιασδήποτε νέες προτάσεις για αλλαγή των ορίων πρέπει να υποστούν την ίδια βάσανο στην οποία υποβάλλουμε και τον αρχικό καθορισμό των ορίων πρέπει να κάνουμε λοιπόν την ίδια απαιτητική διαδικασία. Καλωσορίζω λοιπόν την ε, προσέγγιση της Κομισιόν και τις διάφορες εκθέσεις που έχουν εδώ ε, μπει σε πολύ μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας και αναμένω τις περαιτέρω εξελίξεις στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος ε, βουλευτής θέλει τον λόγο. Κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, λόγω της ε, μεγάλης ποσόστοσης καρκίνου στην Ευρώπη, ε, παράλληλα έλλειψη εκπαίδευσης της κοινωνίας για το κίνδυνο από τις οσίες, πάνε χέρι-χέρι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να απουσιάζει από το θέμα αυτό την εκπαίδευση. Είναι προστασία των εργαζομένων. Είναι τα απαραίτητα που πρέπει να ξέρει και να χρησιμοποιήσει ένας εργαζόμενος. Να υποχρεώνεται ο εργοδότης, το εργοστάσιο, τα συνδικάτα να είναι πλήρης εκπαιδευμένος και εξοπλισμένος ο εργαζόμενος για να προστατέψει την υγεία του. Όταν λείπει αυτή η κουλτούρα, τα, αποτελέσματα είναι φοβερά. Μιλάμε για μεγάλη ποσόστοση καρκίνο από παιδιά έως μεγάλης ηλικία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί τα, τα τελευταία 15-20 χρόνια στην Ευρώπη δεν δίνεται καμία σημασία στην προστασία, στην εργασία. Αυτό είναι η βάση. Από εκεί και πέρα θα φτάσουμε και στο βιομηχανικό κομμάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ ορισμένα, μια που είμαστε τόσο λίγοι. να σας πω την άποψή μου. Έχουμε κάπως διαφορετική άποψη. Τώρα δεν θέλουμε να ξανασχοληθούμε με θέματα που μας έχουν ήδη απασχολήσει. Αυτή είναι μια βασική αρχή. Και ελπίζω να τη συμμερίζονται και οι άλλοι σκιώδεις εισηγητές. Δεύτερον, συμμερίζομαι κάποιες ανησυχίες για κάποιες ουσίες που έχουν παραλυφθεί από, αυτό το δεύτερο, από αυτή τη, τη δεύτερη δέσμη. Όταν εργαζόμεθα επί της, ε, για την πρώτη δέσμη, περιμέναμε ότι θα έχουμε το διπλό αριθμό ουσιών στη δεύτερη δέσμη και ότι θα αντιμετωπιστεί και το θέμα ε, του ντίζελ. Αλλά δεν βλέπω να συμπεριλαμβάνεται. Κατά τη συζήτηση της πρώτης δέσμης, ε, το Κοινοβούλιο δεν πρότεινε οριακές τιμές για πρόσθετες ουσίες, γιατί ακριβώς μας είχατε υποσχεθεί, μας είχε υποθεί δηλαδή, ότι θα γινόταν κάτι περαιτέρω. Άρα θέλουμε να μάθουμε πότε θα συμπεριληφθούν και αυτές οι ουσίες. Πότε θα έχουμε προτάσεις. Τρίτον, για την ε, Φόρμα Αλδείδη ξέρω ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ε, κοινωνικών εταίρων ότι θα πρέπει να υπάρχει δεσμευτικός δεσμευτική οριακή τιμή για επαγγελματική έκθεση και εφόσον υπάρχει συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, πρέπει να τηρηθεί. Αυτή είναι πάντα η προσέγγιση μας. Άρα τίθεται το ερώτημα. Θα τηρηθεί τελικά. Και πότε. Και κάποιες ερωτήσεις τώρα. Και ξέρω ότι θα έχουμε και άλλες ερωτήσεις αργότερα προς την κυρία Επίτροπο και τώρα και μεταγενέστερα βέβαια. Όταν θα έχουμε περισσότερους παρόντες δεν θα έχουν πάει όλοι οι διακοπές. Εντάξει, ίσως έχουν και άλλες ε, δραστηριότητες. Οπότε παρακαλώ. Έχετε το λόγο κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ήμουν ε, μέλος του Κοινοβουλίου και ξέρω ότι οι τελευταίες ε, μέρες πριν τις διακοπές Έχεις πολλά να κάνεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι πολλοί πρέπει να μην είναι, αλλού, να μην είναι εδώ, είναι αλλού και αργότερα μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Τώρα για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Ευχαριστώ την κυρία Μάκιντα για την παρέμβασή της και τις παρατηρήσεις της. Εκτιμώ τις παρατηρήσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει περισσότερη επιστημονική βάση, να έχουμε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και να, να είναι πάντα ο στόχος μας να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στον τόπο εργασίας. Και υπάρχουν και άλλα νομοθετήματα. Αλλά αυτό στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων στον τόπο εργασίας. Άρα πρέπει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα είναι προτεραιότητά μου. Στην ανακοίνωσή μας για την ε, επαγγελματική υγεία και ασφάλεια τονίσαμε ότι θα υπάρξουν διάφορες δέσμες ε, καρκινογόνων ουσιών. Τότε ήταν η παρουσίαση της δεύτερης δέσμης. Όπως είπα και στην ε, παρουσίασή μου, θα υπάρξει και τρίτη δέσμη. Και θα δούμε μήπως χρειαστεί και τέταρτη. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε ουσία που αναφερόταν στον ε, κατάλογο που κατέρτισαν πριν από χρόνια η κοινωνική εταίροι και που θέλει κάποια τώρα ενημέρωση δεν σημαίνει πως δεν ε, ασχολούμεθα με όλες τις ουσίες αλλά προτιμώ να σας υποβάλω τις προτάσεις επί των ουσιών επί των οποίων ε, είμαι θα ήδη έτοιμοι καλύτερα να το κάνουμε σταδιακά σε τρεις-τέσσερις δέσμες Αντί να περιμένουμε μέχρι να έχουμε όλες ε, τις ε, πληροφορίες που θέλουμε για όλες τις ε, ουσίες, γιατί αυτό δεν θα μας επέτρεπε να υποβάλουμε προτάσεις ενδεχομένως πριν το τέλος του 18. Νομίζω ότι είναι καλύτερη αυτή η προσέγγιση, γιατί επιτυχάνουμε περισσότερα μέσω αυτής της διαδικασίας και ταχύτερα. Για την παρέμβαση της κυρίας Κούνεβα. Φυσικά, πρέπει πάντα αυτή να είναι η αντιμετώπιση μας, η προστασία των εργαζομένων. Αν δείτε την ανακοίνωσή μας, ε, που ε, παρουσιάστηκε πριν από δίμηνο περίπου, εκεί ακριβώς εξετάζουμε ποια είναι η συγκεκριμένη πραγματικότητα στους τόπους εργασίας. Και αυτό που έμαθα συζητώντας με πολλούς εκπροσώπους και των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργαζομένων και των ε, εργοδοτών και των μικρομεσαίων ήταν ότι πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία όπως για τις καρκινογόνες, αλλά επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε την εφαρμογή στους τόπους εργασίας, γιατί η εφαρμογή της νομοθεσίας μας είναι πάντα μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό έχουμε απαιτήσει από το φορέα μας στο Μπιλμπάου να εργαστεί από αυτού, να δώσει κατευθυντήρε γραμμές, να βοηθήσει ιδιαίτερα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να εφαρμόσουν την νομοθεσία αυτή, να τους βοηθήσουμε να κάνουν ε, εκτίμηση των κινδύνων γιατί η προστασία κατά των καρκινογόνων δεν είναι μόνο τα όρια αλλά είναι να ε, κάνει ε, η επιχείρηση ό,τι μπορεί να προστατεύσει τους εργαζομένους, να αντικαταστήσει τις ουσίες με άλλες, να εργάζεται σε ένα κλειστό περιβάλλον. Και αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, τότε έχουμε και αυτά τα όρια. Αλλά το βασικό είναι να υπάρχει σωστή προσέγγιση, η σωστή νοοτροπία. Και νομίζω ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχει αυτή η κουλτούρα, αλλά φυσικά μπορούμε πάντα να βελτιώσουμε την κατάσταση και εδώ είμαστε για να τους στηρίξουμε. Και όσοι δεν έχουν αυτή την, νομοθε... Ε, νοοτροπία, η νομοθεσία θα τους βοηθήσει να αλλάξουν ε, νοοτροπία. Δουλεύουμε λοιπόν ε, στα διάφορα επίπεδα και νομοθεσία και εφαρμογή της και κατευθυντήρες γραμμές ο φορέας μας ως μας βοηθάει πολύ και υπάρχουν και άλλες οδηγίες στα πλαίσια του ως και για την κυρία Έλσκοκ για το ποιες ουσίες έχουμε συμπεριλάβει και τι μπορείτε να κάνετε εσείς φυσικά είναι δικό σας θέμα. Είστε συνομοθέτες. Εμείς υποβάλλουμε τις προτάσεις και μετά εσείς οι συνομοθέτες, κοινοβούλιο, συμβούλιο, εσείς ε, καθορίζετε το πώς θα τις αντιμετωπίσετε δεν περιλαμβάνονται όλε οι ουσίε που θα αναμένατε στη δεύτερη δέσμη. Σα είπα ότι αυτό έχει να κάνει με τη διαδικασία. Ε, Έπρεπε να επιλέξουμε ή θα αναβάλαμε την ε, παρουσίαση τη δεύτερη δέσμη για να τι έχουμε όλε, ή θα υποβάλαμε μια δεύτερη δέσμη με όσε ουσίε μπορούμε να υποβάλουμε και παράλληλα συνεχίζουμε να κάνουμε τι αναγκαίε μελέτες και τι συλλογή στοιχείων για να δούμε τι επιπτώσει έχει στον τόπο εργασία για τι υπόλοιπε. Δεν είναι λοιπόν η τελευταία μα πρόταση αυτή θα υπάρξει και μια τρίτη, είναι υποεκπώνηση και νομίζω ότι θα χρειαστεί και τέταρτη. Σας ελπίζω ότι τον... Σας ε, υπόσχομαι ότι τον επόμενο Ιανουάριο του 2018 θα έχουμε την τρίτη δέσμη και θα δούμε για την τέταρτη γιατί εκεί δεν έχουμε καθορίσει καν ε, ποιες ουσίες θα περιλάβει οπότε μπορείτε να μας κάνετε και συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ υπέροχα όλα αυτά ότι θα έχουμε τρίτη και τέταρτη δέσμη και περιμένουμε. Υπάρχει κάποιος ε, βουλευτής που θα θέλει να υποβάλει ερώτηση. Ορίστε. Ο κύριος Χότς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρα. Από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα και ευχαριστούμε τους φιλοξενούμενους μας που ήρθαν εδώ για να συζητήσουμε τους κινδύνους αυτούς. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία και φαίνεται άδικο ότι ασθενούν εργαζόμενοι μόνο και μόνο γιατί πάνε στη δουλειά τους. Είναι σωστό που αυτά τα ζητήματα τα συζητούμε. Έχω μία-δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Μία έγκυος, παραδείγματος χάρη. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τις εγγύους στο κάτω-κάτω εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μικρό ε, ανθρώπινο όν που μπορεί να το βλάψουν οι καρκινογόνες ουσίες και οι μεταλλαξιογόνες ουσίες, να επηρεάσουν το έμβριο. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Αν χρειάζονται δηλαδή ειδικά μέτρα για αυτή την περίπτωση της εγγύους. Δεύτερον, τι γίνεται όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία στο χώρο εργασίας. Ε, θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, κανόνες για την προστασία ανθρώπων με αναπηρία στον τόπο εργασίας, στον χώρο εργασίας. Όχι τόσο για να βρεθούν σε μια προνομιούχο θέση, αλλά να υπάρχει εγγύηση ότι θα προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι από τις καρκινογόνες και τις μεταλλαξιογόνες ουσίες. Για το γενικότερο θέμα των επαγγελματικών ασθενειών και των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών. Όσον αφορά λοιπόν για αυτό το θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κίνδυνος αυτές οι ουσίες που έχουν συγκεκριμένο να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο σε συγκεκριμένες ομάδες ε, ανθρώπων. Η κυρία Τάισον, σας ευχαριστώ για τις εγγύους τους ανθρώπους με αναπηρία αν έχουμε χρειαζόμαστε συγκεκριμένους κανόνες για αυτούς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια προσέγγιση που προστατεύει τους πάντες. Αυτή είναι η υποχρέωση ενός εργοδότη να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται. Και όταν οι έγκυοι εργάζονται και οι ανάπηροι εργάζονται χρειάζεται προστασία. Τώρα χρειαζόμαστε ειδικού κανόνες για αυτούς. Έχω κάποια ιδέα, αλλά πρέπει να πω ότι δεν ξέρω αν έχουμε ε, λεπτομερείς ειδικού κανόνες σε αυτή την νομοθεσία ή αν χρειαζόμαστε ειδικού κανόνες. Χρειάζεται να συμβουλευτώ αυτούς που γνωρίζουν ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Δεν μπορώ έτσι εκ του προχείρου να απαντήσω και να εκφράσω προσωπικές απόψεις. Μπορούμε να το εξετάσουμε το θέμα. Αναφερθήκατε και στα άτομα με αναπηρία. Θα ήθελα να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να επιταχύνει κάπως την έκθεση για την προσβασιμότητα, για την πράξη περί προσβασιμότητας. Δεν σχετίζεται με τις επαγγελματικές ασθένειες, αλλά την πρόσβαση στο χώρο εργασίας. Να είναι πιο εύκολο οι άνθρωποι αυτοί να βρουν δουλειά, να έχουν πρόσβαση στη δουλειά και να ζουν ανεξάρτητοι. Αλλά πολλούς μήνες τώρα ε, συζητούμε αυτή την πρόταση, ίσως και χρόνο. Μήπως κυρία Πρόεδρε μπορείτε να σπρώξετε τους συναδέλφους σας ε, στο Κοινοβούλιο να κινηθούν ταχύτερα, διότι εδώ έχουμε συγκεκριμένους κανόνες, ειδικού κανόνες που χρειαζόμαστε και ελπίζω σύντομα να μπορούμε να δείξουμε στους ανθρώπους με αναπηρία ότι τους φροντίζουμε από όλε τις πλευρές. Τώρα χρειαζόμαστε ειδικέ κατηγορίες, φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν εφικτό. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως μια απευθείας απάντηση τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τάισον. Θα πάμε τώρα στους ομιλητές του πάνελ. Αντρέα Χάρτβικ, από την Επιστημονική Επιτροπή για τα όρια τα επαγγελματικά και τα όρια έκθεσης, Έλκε Σνάιντερ, πρόληψη και έρευνα, η σχετική μονάδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή στον τόπο εργασίας, Λοράν Φούγκαλ, ερευνητής στο ETUC, Ρεμπέκα Σμιθ, σύμβουλος στο τμήμα κοινωνικών υποθέσεων της Business Europe. Θα κάνετε σύντομες εισαγωγές. Από την κυρία Χάρτβικ μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω εδώ και εκ μέρου του ΣΚΟΛ να παρουσιάσω την προσέγγιση μας για την αντιμετώπιση των καρκινογόνων ουσιών. Όπως φαίνεται και στον τίτλο, η Επιστημονική Επιτροπή για, τα, ε, την επαγγελματική έκθεση είναι μια επιστημονική επιτροπή και εν γέννη θα θέλαμε να προτείνουμε ή δυνατόν ε, να δίδονται ε, κάποιες επιστημονικές συμβουλές όσον αφορά τα καρκινογόνα και τα μεταλλαξιογόνα. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, να κάνουμε διάκριση με, μεταξύ καρκινογόνων όσον αφορά τις χαμηλές δόσεις, χαμηλή έκθεση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τα επίπεδα της έκθεσης ευτυχώς έχουν μειωθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια και αυτό που είναι σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε τις καρκινογόνες ουσίες υπό το φως αυτών που συμβαίνουν στα εναπομένοντα επίπεδα εκθέσεως. Προσπαθούμε να κάνουμε αξιολόγηση πληρέστατη των στοιχείων μας, επιδημιολογικά στοιχεία ανθρώπων στον τόπο εργασίας, ε, επίσης στοιχεία για την ε, επίδραση που έχουν οι καρκινογόνες ουσίες στα ζώα και τρόπο που δρούν τα χημικά καρκινογόνα, οι χημικές καρκινογόνες ουσίες. Τι απορρέει από τη μελέτη στην Επιτροπή μας, ε, είτε μπορούμε να προτείνουμε κάποια τιμή με βάση την υγεία, κάποια όρια, μπορώ να σας δώσω αργότερα κάποια παραδείγματα, ή να δώσουμε κάποιες εκτιμήσεις αριθμητικές για την έκθεση, να πούμε σε αυτά τα επίπεδα έκθεσης έχετε αυτό το κίνδυνο που υπολογίζεται βάσει επιστημονικών στοιχείων. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν κατορθώνουμε να δώσουμε κάποια πρόταση συγκεκριμένη, ούτε αριθμητικό ποσοστό ε, κινδύνου όταν έχουμε στοιχεία που δεν μπορούν να μα οδηγήσουν σε συμπέρασμα που καθορίζονται σε ένα επίπεδο, το επίπεδο αυτό είναι πραγματικά ασφαλέ στον τόπο εργασία. Δεν έχουμε αυτή τη σιγουριά. Ε, βλέπουμε εδώ αυτό το γράφημα όσον αφορά τα πειράματα στα ζώα και βλέποντας τα παλιά στοιχεία για την έκθεση έχουμε στοιχεία όσον αφορά τα, τις καρκινογόνες ουσίες και έκθεση σε αυτές τις ουσίες, ε, έκθεση σε υψηλά επίπεδα ή συγκριτικά ψηλά επίπεδα. Πρέπει να δούμε όμως τι γίνεται σε χαμηλά επίπεδα εκθέσεως. Εδώ βλέπετε ε, τις σχέσεις δόσεων ανταπόκρισης. Βλέπουμε μπορεί να υπάρχει γραμμική ανταπόκριση, οπότε μπορείτε να κάνετε προβολή από την έκθεση σε υψηλή δόση, σε χαμηλή δόση, όμως ανάλογα με τον τρόπο δράσης των ουσιών των συστατικών, ίσως η καρκινογόνα δράση γίνεται προφανής μόνο σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Παραδείγματος χάρη, αν έχετε μηχανισμό αντίδρασης που είναι εκτός του DNA, είναι η πράσινη ε, γραμμή στην οθόνη, ή έχετε άλλη, άλλου τύπου σχέση σε χαμηλές δόσεις, χαμηλότερο κίνδυνο από ό,τι θα προβλεπόταν από τα υψηλότερα επίπεδα έκθεσης που βλέπετε με την κίτρινη γραμμή ή με την ανώτερη γραμμή που βλέπετε, την κόκκινη, μπορείτε να έχετε υψηλότερο κίνδυνο ακόμα και με χαμηλή δόση. Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που δρούν οι ουσίες και εξετάζουμε όλα τα στοιχεία. Αν δεν έχουμε στοιχεία, τότε προβλέπουμε μια γραμμική σχέση δόσης ανταπόκρισης. Και αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση, αυτή η γραμμική ανταπόκριση, στις περισσότερες ε, περιπτώσεις. Τώρα, ε, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Κάνουμε διαφοροποίηση ανάλογα με τον τρόπο δράσης. Αν οι καρκινογόνες ουσίες είναι γονιδιοτοξικές ουσίες ή μη γονιδιοτοξικές καρκινογόνες ουσίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι αν έχουμε ένα, μια καρκινογόνη ουσία που επηρεάζει το DNA, μπορεί να προβλέψει κανείς ότι ακόμα και αν έχεις χαμηλά επίπεδα έκθεσης και γίνεται ζημιά στο DNA που ίσως μετατραπεί σε κάποιες μεταλλάξεις, έχεις ακόμα κινδύνους ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα έκθεσης, αλλά δεν μπορείς να καθορίσεις το επίπεδο στο οποίο είσαι πραγματικά ασφαλής και να πεις ότι δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος. Λοιπόν, τι κάνουμε, εξετάζουμε αυτές, αυτά τα συστατικά και βλέπουμε αν έχουμε τα στοιχεία, κάνουμε αξιολόγηση αριθμητική του κινδύνου ή δυνατόν, διαφορετικά δεν δίνουμε κάποια τιμή αν δεν έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία. Λέμε, καλώς είναι καρκινογόνο, άρα η έκθεση πρέπει να είναι όσο πιο χαμηλή γίνεται. Όμως, έχουμε και πολλές καρκινογόνες ουσίες, που ε, οδηγούν σε μια μη γονιδιοτοξική αντίδραση αν αντιρρήσουν με την ε, διέρεση του κιτάρου ή συμβάλλουν σε άλλες διεργασίες που οδηγούν σε καρκινογένεση, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έχεις ένα, ένα αποτέλεσμα ε, που μοιάζει με κάποιο όριο. Μπορεί να έχεις ένα επίπεδο που είσαι ασφαλής. Μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση για αυτές τις ουσίες και ίσως μετά να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για αυτού του για αυτού του είδους την αντίδραση. Προτείνουμε τέσσερις ομάδες ξεχωριστές, δεν είναι σταθερές κατηγορίες. Είναι κάποια ομαδοποίηση, αν θέλετε, να κάνουμε διάκριση μεταξύ τρόπων δράσεως. Πρώτα απ' όλα έχουμε γονιδιοτοξικές καρκινογόνες ουσίες, όπου έχουμε εναπομένοντα κίνδυνο ακόμα και σε πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης. Β, είναι μια ουσία όπου δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, αλλά θεωρούμε ότι ανήκει, είναι παρόμοια δράση με την ομάδα Α στην D έχουμε ένα μηχανισμό που πραγματικά προβλέπουμε ένα όριο και στην ομάδα C μπορούμε να πούμε ότι πιθανότατα υπάρχει ένα πρακτικό κατώτατο όριο που μπορούμε να προτείνουμε με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε για το πώς επηρεάζεται η υγεία. Αυτή λοιπόν είναι η γενική μας ε, προσέγγιση στην περίπτωση γονιδιοτοξικών καρκινογόνων, ομάδα Α και Β, πολύ συχνά μπορεί να μην είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα χαμηλότερο όριο έκθεσης βάση ε, στοιχείων για την υγεία. Αν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία μπορούμε να κάνουμε ξελόγηση του κινδύνου βάσει ε, γραμμικής προβολής από τα δεδομένα επίπεδα έκθεσης ανθρώπων και ζώων και τα αποτελέσματα που έχει αυτή. Στην περίπτωση έμεσης δράσης, λέμε καλώς μπορούμε να εντάξουμε τις ουσίες στην κατηγορία D αν έχουμε πραγματικό όριο που μπορεί να καθοριστεί ή στην ομάδα C που προβλέπουμε ότι έχουμε κάποια επίπεδα έκθεσης κάτω από τα οποία η καρκινογόνα δράση δεν μας αφορά πλέον. Σε όσες περιπτώσεις εξετάζουμε κατά πόσο υπάρχει κάποιος βιολογικός επηρεασμό και εξετάζουμε και επιδημιολογικά στοιχεία, τα προτιμούμε. Αν έχουμε στοιχεία για τους ανθρώπους για κάποια κακινογόνα ουσία. Αυτές είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες. βάλουμε υπόψη και τα στοιχεία τα πειράματα στα ζώα και διάφορα μηχανιστικά στοιχεία που έχουν ε, δημοσιευθεί στα διάφορα επιστημονικά συγγράμματα για να μπορούμε να δούμε ποια ε, είναι οι σχέσεις ε, έκθεσης, αντίδρασης στα πολύ, στα πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα ήθελα. Λίγο πίσω μπορούμε να πάμε στις διαφάνειες σας παρακαλώ. Μία πίσω. Ένα παράδειγμα είναι το χρώμιο 6. Είναι καρκινογόνο στα, στους ανθρώπους και στα ζώα στο περάτημα. Είναι γονιδιοτοξικό, μεταλλαξιογόνο, καρκινογόνο. Ε, οπότε προβλέπουμε γραμμική σχέση δόσης αποτελεσμάτων παρόλο που ίσως μειώνεται κάπως το χρώμιο 6 στο σώμα, το βάζουμε στην ομάδα 1 αυτή την ουσία και οι, αξ... τιμές κινδύνου βασίζονται στη γραμμική προβολή για τον καρκίνο του πνεύμονα. άλλα μέταλλα, νικέλιο και κάδμιο, και αυτά είναι καρκινογόνα για τους ανθρώπους και στα πειραματικά ζώα, στα ζώα των πειραμάτων, έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης, δεν είναι άμεσα αγωνιδιοτοξικές ουσίες, διότι παρεμβαίνουν στη διαδικασία επισκευής του DNA. Άρα δεν είναι άμεση αντίδραση με το DNA, αλλά επηρεάζονται οι πρωτεΐνες. Άρα μπορεί να προβλέψουμε πρακτικά κατώτατα όρια, όμως Μιλώντας για τα καρκινογόνα, προβλέπουμε ότι τα ίδια συστατικά ίσως να έχουν και μη καρκινογόνα αποτελέσματα. Και για τα δύο μετάλλα, και για το νικέλιο και για το κάδμιο. Και αυτό σε πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης. Επίσης, στην περίπτωση του νικελίου μπορεί να οδηγήσουν στην τοξικότητα του πνεύμονα, στην περίπτωση του καδμίου, τοξικότητα στα νεφρά. Οποιαδήποτε τιμή προτείνουμε θα πρέπει να προστατεύει όχι μόνο από ε, καρκινογόνες συνέπειες αλλά άλλες τοξικές συνέπειες και γι' αυτό προτείνουμε μια τιμή που προστατεύει από, την, από τοξικές συνέπειες τα όργανα και ε, καρκινογόνες συνέπειες. Προσπαθούμε να συναθρήσουμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία, να δώσουμε συμβουλές, δεν καθορίζουμε τιμές, απλώς προτείνουμε κάποιες τιμές, διότι Πώ υλοποιούνται οι μελέτε, πώς μεταφράζονται σε κινδύνους στον τόπο εργασία δεν είναι εύκολο. Ε, κάνουμε την καλύτερη πρόταση για την προστασία των εργαζομένων σε, μια συγκεκριμένη, ε, σε συγκεκριμένο τόπο εργασία αυτή τη ουσία. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Σνάιντερ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στην Εργασία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Επιτροπής που μας κάλεσε και πάλι για να παρουσιάσουμε την δουλειά μας. Θα ήθελα να προσθέσω στην νομική και την επιστημονική πτυχή πέρα από τα όρια έκθεσης την πτυχή του χώρου εργασίας. Δεν θα αναφέρω όλα τα στοιχεία που έχω, τα έχετε ξαναδεί. Ε, σε δύο μηνύματα θα αναφερθώ. Μάλλον έχετε ακούσει τον αριθμό του 4 έως 8% των θανάτων στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με τα καρκινογόνα στην δουλειά. Θεωρούμε όμως ότι όταν εξετάζουμε αυτά τα νούμερα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι διαφέρουν ε, κατά πολύ αναουσία και είναι πολύ ψηλότερα για έκθεση σε κάποιες από τις ουσίες. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι πολλές από αυτές τις ουσίες έχουν ταυτοποιηθεί μέσω έκθεσης ε, στους ε, εργαζόμενους, ειδικά των εργαζομένων που είναι πολύ εκτεθειμένοι. Μια χαρακτηριστική ουσία, παραδείγματος χάρη, είναι ο αμύαντος. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι εργαζόμενοι συχνά εκτίθενται σε πολλές καρκινογόνες ουσίες ε, ταυτοχρόνως. Ε, παραδείγματο χάρη εδώ πέρα έχουμε 7 ουσίες. Η πρώτη ομάδα εργαζομένων που αναφέρονται εδώ, μηχανικοί, συγκολητέ, ε, παραδείγματο χάρη, εκτίθενται σε δύο ουσίες ήδη, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλεα. Οπότε εκτίθενται σε πολλές καρκινογόνες ουσίες οι εργαζόμενοι ταυτόχρονα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, αλλά και για όσους δουλεύουν σε υπηρεσίες, π.χ. κομμότριες, κομμωτές που εκτίθενται σε διαλυτικές ουσίες ή και σε εμπογές που είναι καρκινογόνες. Ακούσαμε την αξιολόγηση αντικτύπου και του, του ωφέλου στην υγεία. Η προηγούμενη ομιλήτρια είπε πως ε, υπάρχουν και άλλες ιδιότητες των καρκινογόνων ουσιών. Ε, συνήθως οι καρκινογόνες ουσίες έχουν πολλές επιδράσεις. Π.χ. υπάρχει συχνά μια ευαισθητοποίηση, έχω βάλει εδώ πέρα π.χ. τα ροκανίδια, τα οποία επηρεάζουν το αναπνευστικό, την ε, επιδερμίδα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν και μία υπερευαισθησία. Άλλες προτάσεις είναι παρόμοιες, ε, μπορεί να είναι ε, π.χ. τοξικές ουσίες, είτε αν καταποθούν, είτε αν τις εισπνεύσει κανείς, είτε μέσω της επαφής με το δέρμα, αλλά προκαλούν ερεθισμό, άλλα μπορεί να αποκαλούν ναυτία και κίνδυνο ατυχήματος. Τι θέλω να πω εδώ. Τα πιθανά ωφέλη πέρα από τις, τα ζητήματα διοντολογίας και ηθικής ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλα και άρα έχουμε ένα ζήτημα πολύ ευρύτερο από το κόστος ε, ή την αποφυγή του κίνδυνου καρκίνου. Παραδείγματος χάρη μια υπερβεστησία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της εργασίας και το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος το απευθείας ε, της έκθεσης στο καρκινογόνο. Οπότε το οικονομικό όφελος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από το να εξετάζουμε μόνο την πτυχή του καρκίνου. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάποια αποτελέσματα από δύο από τις ε, δημοσιεύσεις μας, παρότι ήταν μια έρευνα που έγινε μεταξύ των κρατών μελών για το πώς αντιμετωπίζουν τα όρια έκθεσης για τα καρκινογόνα και το δεύτερο είναι μια έκθεση που εξετάζει τις μεθόδους αξιολόγησης για έκθεση και αρρώστιες και τις εθνικές πολιτικές που σχετίζονται με τις καρκινογόνες ουσίες. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, της δεύτερης έκθεσης, κάποια από τα ευρήματα που έχουμε είναι ότι συχνά στα δεδομένα που έχουμε π.χ. για την αξιολόγηση αντικτύπου δεν καλύπτονται οι τομείς των υπηρεσιών. Επίσης, έχει ήδη αναφερθεί ο κίνδυνος των ευπαθών εργαζομένων που εκτίθενται και μπορεί να εκτίθενται και να μην αξιολογείται αυτό. Μπορεί να μην υπάρχουν στα δεδομένα κάποιες ομάδες και έχουμε μια πιθανή υποεκτίμηση των αποτελεσμάτων. Επίσης θα πρέπει να δούμε ε, το ότι δεν υπάρχουν στρατηγικές επιστροφής στην εργασία για όσους αρρωστήσουν από καρκίνο και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, κοιτώντας τα αποτελέσματα της έκθεσης θα ήθελα να τονίσω την σημασία των ουσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια διαδικασιών και επηρεάζουν πολλούς εργαζόμενους. Τις 7 ουσίες ε, τους ε, έχουμε τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που είναι ένα μείγμα που παράγεται προκύπτει. Φυσικά είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί γιατί συχνά είναι το αποτέλεσμα της καύσης ε, και δεν είναι εύκολο να αποφευχθεί, οπότε επιλέγουμε εδώ πέρα μία ουσία ως την κύρια ουσία για τις ε, μετρήσεις ε, και ε, εξετάζουμε διάφορες ομάδες κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητε, αλλά αν δούμε άλλες έρευνες και από την Αυστραλία και τον Καναδά βλέπουμε ότι αφορά και άλλους εργαζόμενους, π.χ. τους αγρότες, όσους δουλεύουν στην κουζίνα εστιατορίων, αλλά και ε, όσους δουλεύουν στο ΕΚΑΒ, πυροσβέστες ε, και λοιπούς. Π.χ. υπάρχει και ε, καπνός που παράγεται στα χειρουργεία, που μοιάζει πάρα πολύ με τον καπνό που παράγεται όταν κόβουμε κάτι με λέιζερ. Και εκεί παράγονται και αρωματικοί υδρογονάνθρακες και δεν υπάρχει πρόληψη. Δηλαδή όταν κόβουμε κάτι με λέιζερ μπορεί να υπάρχουν περισσότερα μέτρα πρόληψης στη βιομηχανία παρά στα χειρουργεία, όπου η έκθεση είναι παρόμοια και υπάρχει λιγότερη πρόληψη στα χειρουργεία. Όσον αφορά τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια αξιολόγηση της επιδερμίδας για να αποφευχθεί η απορρόφηση αυτών των ουσιών. Η αξιολόγηση λοιπόν της κατάστασης επιδερμίδας είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δεύτερο έβριμα της έκθεσης αυτής. Εξετάσαμε το πώς καλύπτονται οι ευπαθείς ομάδες από τη συλλογή των δεδομένων και βλέπουμε ότι ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών αλλά και για κάποιες ομάδες όπως οι νεαροί εργαζόμενοι. Ε, δεν υπάρχουν ε, λεπτομέρειες γιατί συχνά οι νεαροί ε, δουλεύουν με προσωρινές συμβάσεις και λαμβάνουν καθήκοντα όπως η συντήρηση και λόγω της έλλειψης εμπειρίας συχνά είναι και στη δουλειά εκείνη η οποία απαιτεί λιγότερα προσόντα. Όμω οι μελέτε δείχνουν ότι οι νεαροί μπορεί να είναι πιο εκτεθειμένοι στι καρκινογόνε ουσίε για τον ίδιο ακριβώ λόγο και να εκτίθενται σε πολλές ε, καρκινογόνες ουσίες ε, ταυτόχρονα. Ε, ίσως και περισσότερο από τον μέσο εργαζόμενο. Είναι σημαντικό μήνυμα αυτό γιατί οι νεαροί εκτίθενται και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τους άλλους και εάν δούμε ειδικά τους εκπαιδευόμενους, τους βοηθούς, ειδικά σε χειρονακτικές εργασίες, π.χ. στα κομμωτήρια, υπάρχει διαφορά και αντικτύπωση και όμως δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για να αξιολογήσουμε την κατάσταση όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα ήθελα τώρα να έρθω στην δεύτερη έκθεση για τα όρια έκθεση στο χώρο εργασίας στα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο βλέπουμε από αυτή την έκθεση, η έκθεση αυτή είναι κάπως παλιά, αλλά υπάρχουν ε, πέρα από τα νούμερα και κάποιες γενικές δηλώσεις. Εκεί υπάρχει ένας αριθμός ορίων που ποικίλει ε, ανά μέλος και χρειάζεται πολλής χρόνος μέχρι να τεθεί ένα όριο. Πολλά κράτη-μέλη αναφέρουν ότι έχουν υιοθετήσει τις τιμές από άλλες χώρες ε, και έτσι υπάρχει δυνατότητα να μοιραζόμαστε πληροφορίες και έρευνα μεταξύ κρατών μελών. Οι συχνότερες δυσκολίες είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για την έκθεση ή τοξικολογικά δεδομένα και βεβαίως προβλήματα όσον αφορά την επίτευξη μιας συνένεσης. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει προσθέμενη αξία το να μπει ένα όριο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να καταλήξω με λίγα λόγια για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το θέμα της σημερινής ακρόασης. Το πρώτο είναι μία μελέτη σκοπιμότητας ε, που κάναμε για να δούμε αν μπορούμε να συμπληρώσουμε τα δεδομένα με μία έρευνα για την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες και σε άλλους παράγοντες. Ε, λάβαμε μόλις χτες την έκθεση με κάποιες συστάσεις για την πιθανή αλλαγή μεθοδολογίας όπως αυτή που χρησιμοποιείται στην Αυστραλία και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για το αν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οπωσδήποτε κάτι τέτοιο θα συνεισέφερε στο να έχουμε καλύτερα δεδομένα για το πώς εργαζόμενοι εκτίθενται, σε ποιο βαθμό και ποιες ε, ομάδες εργαζομένων. Η δεύτερη πρωτοβουλία που θα ήθελα να αναφέρω είναι η εκστρατεία για τους υγιείς χώρους εκστρατείας, ε, εργασίας με συγχωρείτε, για το 2018 και 2019. Έχουμε λοιπόν τα εξή θέματα που είναι σημαντικά για τη σημερινή μας συζήτηση. Το ένα είναι ακριβώς τα μηνύματα αυτά για την αξιολόγηση, για την μείωση σε έκθεση σε καρκίνογον στον χώρο εξτατείας και το δεύτερο είναι η προστασία των εργαζομένων με συγκεκριμένες ανάγκες και υψηλότερους κινδύνους είτε επειδή ε, για λόγους ε, της ε, ανατομίας τους ε, είναι πιο ευπαθής είτε για λόγους της έκθεσης, τη, λόγω του είδους της εργασίας ή της έλλειψης ενημέρωσης. Ε, υπάρχει όμως και η διάσταση του φύλου, γιατί κατά κανόνα, όπως είπα, στον τομέα των υπηρεσιών υπάρχει λιγότερη ενημέρωση, ανέφερα τον τομέα αυτών και τον τομέα της υγείας, αλλά υπάρχουν και οι μάγειροι στις κουζίνες με τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες τα ζητήματα είναι τα ίδια. Η απαγωγή αέρα και η αποφυγή έκθεσης ε, του δέρματος. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφέρω την στήριξή μας στον οδικό χάρτη για τις καρκινογονωσίες, μια πρωτοβουλία της Ολλανδικής ε, Προεδρίας για να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης που συνεχίστηκε και μέχρι την Αυστριακή Προεδρία. Θα οργανώσουμε λοιπόν μια ετήσια εκδήλωση και θα προετοιμάσουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο. Η εκδήλωση φέτος θα γίνει στην σχετική έκθεση για την ασφάλεια και την υγιεινή στον χώρο εργασίας και έχουμε τα κράτη-μέλη που θα παρουσιάζουν τις εκστρατείες για τις καρκινογονησίες, το τι κάνουν πρακτικά θα γίνει και μια παρουσίαση από την Ολλανδία για τις συζητήσει που είχαν με τις εταιρείε για την υποκατάσταση ουσιών και έναν οδηγό που είχε συντάξει η σχετική ε, επιτροπή για την ε, έκθεση στην Λοιπόν, επ' ευκαιρία δε της Παγκόσμιας ημέρας καρκίνου δημοσίευσαμε μία έκθεση για το θέμα της ε, επανόδου στην δουλειά μετά από τον καρκίνο. Έχουμε και την ομάδα των Ευρωβουλευτών κατά του καρκίνου και συζητάμε τα αποτελέσματα της περαιτέρω έρευνας ε, μερικών περιπτώσεων συγκεκριμένων εταιριών που συζητάμε και με άτομα που στηρίζουν την επιστροφή στην εργασία μετά από τον καρκίνο. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω εδώ και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ ο κύριος Φόγγελ που είναι ανώτερος ερευνητής στο, της ε, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων. Σας παρακαλώ να μην περιμένετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Είμαι εκπρόσωπο τη ε, Ευρωπαϊκή Νομοσπονδία Συνδικάτων και το πρώτο που να πω είναι ότι ο συμβασμό που επετεύχθηκε την πρώτη δέσμη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου για τη βελτίωση τη ε, προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο. Και το Κοινοβούλιο έπαιξε κινητήριο ρόλο για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματο Επετεύχθη ε, ευρεία πλειοψηφία, 85% υπερψήφισαν τις τροπολογίες που ήταν η βάση του συμβασμού. Νομίζω λοιπόν ότι η προσπάθεια του Κοινοβουλίου να υπάρξει φιλόδοξη νομοθεσία για να προστατεύει τους εργαζόμενους ήδη είχε αποτελέσματα. Και ελπίζουμε και για τις επόμενες δέσμες να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Δεν θα αναφέρω όλα τα ζητήματα που έχει παρουσίασή μου. Θεωρώ ότι αυτό που έχει σημασία είναι κυρίως να καταλαβαίνουμε ότι όταν εγκρίνουμε μία, ένα νομοθέτημα προστασίας των εργαζομένων από τις καρκινογόνες ουσίες πρέπει να σεβόμεθα τις διατάξεις των συνδικών που λένε ότι πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασία των εργαζομένων από όλους τους παράγοντες που μπορούν να τους θίξουν. Για να αποφύγουμε λοιπόν να υπάρξουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην περίπτωση των εργαζομένων. Δηλαδή για τους εργαζόμενους, για παράδειγμα, δεχόμεθα να εκτίθεται σε κινδύνους πολύ μεγαλύτερους από τους κινδύνους που θα θεωρούν το αποδεκτή για άλλα θέματα νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα για την ασφάλεια των τροφίμων, για την εισαγωγή στην αγορά χημικών ουσιών. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχει το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και για την υγεία και προστασία των εργαζομένων υπάρχει σε άλλους τομείς. Τώρα για τη συγκεκριμένη πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή, τη δεύτερη δέσμη δηλαδή, για την ε, αναθεώρηση της οδηγίας για τις καρκινογόνες ουσίες, προτείνουμε μια σειρά από που αφορούν το παράρτημα 1 και το παράρτημα 3 της οδηγίας. Τι ρόλο έχει το παράρτημα 1 είναι ένας κατάλογος διαδικασιών που μπορούν να εκθέσουν τους εργαζόμενους σε κίνδυνο καρκίνου. Και τι είναι διαδικασίες. Δεν είναι απλώς οι ουσίες που κυκλοφορούν, αλλά πρόκειται για μια σειρά από βιομηχανικές δραστηριότητες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνη έκθεση που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Το παράρτημα είναι σημαντικό γιατί καθορίζει για τις διαδικασίες αυτές τον τομέα εφαρμογής της ε, οδηγίας. Αντίθετα με τις ουσίες, εάν θεωρούνται καρκινογόνες, αυτόματα είναι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αν ακόμη δεν έχει ε, κατηγοριοποιηθεί ως καρκινογόνος αλλά ε, πληρεί κάποια κριτήρια και πάλι αυτόματα εντάσσεται. Ενώ για τις διαδικασίες τίποτα δεν εντάσσεται αυτόματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν το παράρτημα 1. Και αυτό το παράρτημα 1 πρέπει να καλύψει τις περισσότερες καταστάσεις που προκύπτουν πραγματικά στην πραγματικότητα στους τόπους εργασίας, στο χώρο εργασίας. Γι' αυτό καλούμε την Κομισιόν να αξιοποιήσει ένα κείμενο που υπάρχει ήδη, ένα κατάλογο που διαμορφώθηκε από τις Ολλανδικές Αρχές, το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας ε, της Ολλανδίας, RIVM, ε, εκεί περιέχεται ένας κατάλογος διαδικασιών και υπάρχει και ο κατάλογος ε, των συνδικάτων. Και αν τις ε, συγκρίνετε αυτές δύο λίστες θα δείτε ότι είναι περίπου ταυτόσιμες. Για να καλύψουμε λοιπόν τις περισσότερες δυνατότητες έκθεσης στην πράξη είναι σημαντικό να μπει στο παράρτημα 1 η εκπομπή από τους κινητήρες diesel γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό ε, στους χώρους εργασίας. Θα επανέλθω. Πρέπει επίσης να καλύψουμε τη σκόνη και τους καπνούς από το, τα ελαστικά, από το καουτσούκ και επίσης πρέπει να συμπεριληφθούν μια σειρά καταστάσεις έκθεσης σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Ανασχοληθούμε με τις εκπομπές από τους κινητήρες diesel. Γιατί πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα ένα αυτές τις διαδικασίες, πρώτα απ' όλα γιατί προκαλούν καρκίνο, υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση, το Διεθνές Κέντρο Ερευνών κατά το, Έρευνας κατά του καρκίνου το έχει τεκμηριώσει και προκύπτουν πολύ συχνά αυτές οι εκπομπές και αυτό σοβαρός λόγος και να δούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ε, μελέτη αντικτύπου, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε σε 60 χρόνια 230.000 θανάτους. Είναι λοιπόν σημαντικός αυτός ο κίνδυνος. Πριν από μερικού χρόνου ε, ε, προέβλεπε η Κομισιόν να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώ τελικά δεν συμπεριελήφθησαν στη δεύτερη δέσμη αυτέ οι εκπομπέ. Προβλήθηκαν διάφοροι λόγοι, αλλά δεν είναι επιστημονικοί. Δηλαδή υπήρξαν πιέσεις. Που στόχο είχαν να δημιουργήσουν αμφιβολίες για την κατάσταση αυτή. Και κυρίως στο να γίνει μια αντιπαράθεση μεταξύ των ε, παλαιότερων και των πιο πρόσφατων κινητήρων. Αλλά δεν ε, είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη τέτοιο κριτήριο. Η οδηγία αυτή δεν αφορά τον εργασιακό εξοπλισμό, αφορά την έκθεση. Άρα αυτή η διάκριση δεν έχει λόγο να υπάρχει. Στην ε, γνωμοδότηση του ΣΚΟΛ που εγκρίθηκε τον ε, Σεπτέμβριο του 2016 με βάση μια μελέτη που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ καταλήγουν σε αποτελέσματα που δεν ισχύουν γιατί οι προϋποθέσεις αυτές, αυτής της μελέτης των ΗΠΑ είναι πολύ διαφορετικές. Στην μελέτη αυτή τα ε, πειραματόζα εξετέθησαν σε, τέσσερις, ε, σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα ε, προστασίας. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα των εργαζομένων σε χώρους όπου παράγονται τέτοιες εκπομπές. Η μελέτη η άλλη αφορά τα τους κινητήρες δίζελ των αυτοκινήτων, τους πιο πρόσφατους. Για το παράδειγμα 3. Πρέπει κυρίως να σκεφτούμε τι κριτήρια θα ορίσουμε για να ορίσουμε μετά τις οριακές τιμές. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να καλύπτουμε την πλειονότητα των πραγματικών καταστάσεων και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Επιμένω επ' αυτού. Αν λάβουμε υπόψη αυτά τα κριτήρια, να ελέγξουμε και τις εκπομπές, συγγνώμη, τις καταστάσεις στις οποίες εκτίθενται οι εργαζόμενες, θα δούμε τότε ότι υπάρχει έκθεση σε διάφορες ουσίες όπως η φορμαντέιδη. Ο στόχος των οριακών τιμών είναι να μειωθούν οι σημερινές οριακές τιμές. Οι τιμές πραγματικής έκθεσης. Για πολλές χώρες υπάρχουν ήδη τέτοιες οριακές τιμές, ανώτατα όρια που έχουν οριστεί μόνο μερός. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πύρα αυτών των χωρών για να καθορίσουμε τις ευρωπαϊκές ανώτατες τιμές. Και πρέπει να είμαστε συνεπείς και με άλλα ευρωπαϊκά νομοθετήματα. Γιατί έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να καθορίσουμε καλύτερες ανώτατες τιμές. Και πρέπει να είμαστε συνεπείς και με το επίπεδο του εναπομένοντος κινδύνου. Δεν είναι δυνατόν για μια ουσία να υπάρχει πολύ ψηλό επίπεδο προστασίας, ενώ για μια άλλη ουσία δεν είναι δυνατόν να είναι σχετικά χαμηλό το επίπεδο προστασίας. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με διαφανή τρόπο. Γι' αυτό στηρίζουμε το αίτημα του Κοινοβουλίου να υπάρξει μία νέα στήλη στο παράρτημα 3 που να αναφέρει τον ε, εναπομένοντα κίνδυνο. Έχουμε λοιπόν πέντε προτάσεις. Δεν θα τις παρουσιάσω αναλυτικά, αλλά είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε περαιτέρω εξηγήσεις. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τρεις ουσίες για τις οποίες δεν έχει καθορίσει η Κομισιόν εκπομπές, μεταξύ των οποίων και η Φορμαλδεΐδη και δύο ουσίες για τις οποίες θέλουμε οι τιμές που προτείνει η Κομισιόν να μειωθούν. Παράδειγμα, τριχλωρεθυλένιο. Η Κομισιόν προτείνει 550 μιλιγράμμ ανά κυβικό μέτρο, όμως βλέπουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτή την ουσία περιορίζουν την έκθεση σε 3 έως 5 mg. Πολύ χαμηλότερε τιμέ από αυτέ που προτείνει το παράρτημα 3. Δεν αναφέρθηκα πολύ αναλυτικά σε όλε τι τροπολογίες. Νομίζω ότι θα τα δούμε στο μέλλον με τον εισηγητή και του σκιώδες του Κοινοβουλίου. Κυρίω προσπάθησα να καθορίσω τα κριτήρια βάσει των οποίων θα υποβάλουμε συγκεκριμένε προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρεμπέκα Σμιθ έχει το λόγο, σύμβουλος στο τμήμα κοινωνικών υποθέσεων της Business Europe. Έχετε το λόγο, κυρία Σμιθ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση που μου κάνατε να έρθω σήμερα. Έτσι οι κοινωνικοί εταίροι θα εκφράσουν τις ε, απόψεις τους. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε τις διάφορες απόψεις εργοδοτών και εργαζομένων έγινε πρώτη, για την πρώτη δέσμη ακρόαση, δέσμη μέτρων για την οδηγία και η πανέμβασή μου θα μοιάζει με αυτήν που έκανα για, την, ε, το πρώτο, πρώτη δέσμη αναθεωρήσεων. Ε, εν γέννη υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρότασή της για τη δεύτερη δέσμη των μέτρων και εν γέννη υποστηρίζουμε τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό να γίνει ένα θεώρηση οδηγίας για τις καρκινογόνες ουσίες, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι καλύπτουμε όλες τις ουσίες που θα πρέπει να καλύπτονται από την ε, οδηγία. Καλωσορίζουμε και το ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδράζεται επί της νομοδοτήσεως της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια, όπου εκεί πετεύχθη συνένεση μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων και κυβερνήσεων και από τα 28 κράτη-μέλη και βέβαια αυτό βασιζόταν σε επιστημονικές συστάσεις του ΣΚΟΛ. Ε, παρόλο που καταλήξαμε σε γενική συνένεση, ίσως κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, θα ακούσει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε συνεργαστεί με την ETUC μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής και καταλήξαμε σε μια γενική συμφωνία επί των ορικό, οριακών τιμών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτές οι οριακές τιμές που συμπεριλήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της, ε, των ε, κατευθύνσεων Βουλευτικής Επιτροπής να εφαρμοστούν. Όλες οι ουσίες που εξετάστηκαν δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη δεύτερη δέσμη αναθεωρήσεων τα συνδικάτα είπαν ότι θα συμπεριληφθούν και άλλες ουσίες σε αυτή τη δέσμη, σε αυτή τη φάση. Πιστεύουμε ότι η επιλογή που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ορθή σε αυτή τη φάση, διότι κατά την άποψή μας είναι σημαντικότατο το εξή. Οποιεδήποτε προτάσεις γίνονται για συμπερίληψη νέων ουσιών ή νέων οριακών τιμών στην οδηγία θα πρέπει να βασίζονται σε αποδεδειγμένα επιστημονικά στοιχεία και αυτές οι ουσίες θα πρέπει να ταξινομούνται ως καρκινογόνες να μην συμπεριλαμβάνονται αυθαίρετα ουσίες στην οδηγία και αυτές οι ουσίες θα πρέπει να έχουν υποστεί την κοινωνικο-οικονομική ανάλυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με αυτό που ήδη αναφέρθηκε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και των οριακών τιμών από τους εργοδότες, αυτές οι οριακές τιμές να είναι προσμετρήσιμες και οι τεχνικές μετρήσεως της έκθεσης να υπάρχουν. Και γι' αυτό εδώ έχουμε κάποια προβλήματα. Όπως ήδη αναφέρθηκε κάποιες από τις ουσίες, όπως είπε η κυρία Επίτροπος, δεν έχουν συμπεριληφθεί ε, ακόμα σε, αυτή τη, αυτό τη δέσμη μέτρων, γιατί χρειάζεται δουλειά. Και είναι καθοδόν και τρίτη δέσμη από ό,τι ακούσαμε και ενδεχομένως και τέταρτη δέσμη αναθεωρήσεων των ουσιών. Καλούμε λοιπόν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τους άλλους εμπλεκομένους φορείς στις εργασίες που θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία να τιμήσουν τη συνένεση που επετεύχθη στη Συμβουλευτική Επιτροπή και να προχωρήσουμε γρήγορα με αυτή την πρόταση. Θεωρούμε ότι είναι μια φιλόδοξη πρόταση και λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα κείμενα, κύματα συγγνώμη, που επίκενται είναι σημαντικό σε αυτή την οδηγία μην καθορίζουμε μόνο οριακέ τιμέ, αλλά να προβλέπονται γενικέ υποχρεώσει του εργοδότε όσον αφορά τη γενική προστασία και τα συναφή μέτρα στον τόπο εργασία. Οι οριακέ τιμέ είναι σημαντικέ, αλλά όλο αυτό πρέπει να εξεταστεί στο γενικότερο πλαίσιο τη ε, οδηγία. Δεν αφορά μόνο τον καθορισμό οριακών τιμών. Συμφωνούμε μεν ότι πρέπει να προσθεθούν αυτέ στην ε, οδηγία, Όμω δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι εργοδότε κάνουν πολύ περισσότερα υποστατεύσει του εργαζόμενου του τομέα, διότι είναι νομικώ υποχρεωμένοι. Εξετάζοντα την ε, νομοθετική διαδικασία, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα ακούσουν απόψει κάποιων εταιριών. Θα πούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίε ε, όσον αφορά την ε, συμμόρφωσή τους με τις οριακές τιμές. Το γνωρίζουμε αυτό και όπως ήδη ε, γνωρίζετε και έχετε ακούσει από τις απόψεις συνδικάτων ότι θα πρέπει να καθοριστούν σε κάποιες περιπτώσεις χαμηλότερες οριακές τιμές. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι έχει βρεθεί στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστή ισορροπία. Βέβαια πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε ότι υπερβάλλεται όσον αφορά τον κατάλογο, άλλοι ότι δεν προχωρήσετε αρκετά. Όμως επετέφθη μια συνένεση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στη Συμβουλευτική Επιτροπή και η ισορροπία που πετέχθη εκεί είναι καλή και ελπίζουμε να διαφυλαχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Κάποιο σχόλιο όσον αφορά το πρώτο κύμα των διαφόρων αλλαγών. Ε, θα πρέπει να επικυρωθεί όλη η προσπάθεια και από το Συμβούλιο. Είμαστε ικανοποιημένοι βέβαια που καταφέρατε να συμφιλιώσετε τις διάφορες απόψεις και να καταλήξετε σε αυτό που θεωρούμε από πλευράς ε, εργοδοτών ε, σαν κάτι αποδεκτό. Είναι αποδεκτός ο συμβιβασμός, χρειάστηκε χρόνος για την τελική συμφωνία. Για μας, τι να σα πω, στην αρχή θεωρούσαμε ότι δεν ήταν ξεκάθαρο θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Υπήρχαν πολλές αποκλίνουσες απόψεις και ανησυχήσαμε ότι ίσως δεν θα προχωρούσαμε. Άρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι τώρα έχει επιτευχθεί μια συμφωνία και ελπίζουμε ότι όσον αφορά αυτό το δεύτερο κύμα ε, και τα μελλοντικά κύματα ε, θα έχουμε αποτελεσματική διαδικασία και θα πετύχουμε συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου το ταχύτερο δυνατόν. Να πω βέβαια ότι υπάρχουν και γενικότερα θέματα που πιστεύουμε ότι καλύφθηκαν με το πρώτο κύμα των ε, τρόπων διαφόρων τοξινών και νομίζουμε ότι αφού λύθηκε το θέμα δεν πρέπει να επαναληφθούν οι συζητήσεις στο δεύτερο τρίτο κύμα των μεταρρυθμίσεων. Επίσης, να πω ότι σαν εργοδότες, επειδή το θέμα συζητείται εκτενέστερα για τις λιποτοξίνες, θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η παρούσα κατάσταση και αν άλλαξε τα τελευταία χρόνια για να καταλάβουμε καλύτερα τι μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε στον τομέα. Κάτι άλλο που αφορά τη Συμβουλευτική Επιτροπή εν γέννη. Ακούστηκαν κάποιες επικρίσεις. Οι επικρίσεις αφορούσαν τον τρόπο που εργάζεται και η Συμβουλευτική Επιτροπή και η Επιτροπή Σκόλο, ότι χρειάζεται πολύ χρόνο για να καταλήξει οριακέ τιμέ και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Δράτω με τι ευκαιρίε να πω ότι τώρα βλέπουμε ότι το έργο της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινούνται όλοι πολύ πιο γρήγορα. Έχουμε σειρά συστάσεων από τη ΣΚΟΛ και συνομιλώντας με συναδέλφους που είχαν συμμετάσχει στην στην ομάδα εργασίας για τα χημικά, ή χημικές ουσίες στη Συμβουλευτική Επιτροπή ότι προσπαθούν να καταλήξουν σε ε, πορίσματα για διάφορες ουσίες, σε φάσμα και αν θέλουμε να κινηθούν πιο γρήγορα αποδεικνύεται ότι αυτό επιτυγχάνεται και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικότατο αυτές οι διαδικασίες ε, ε, διέλευση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή που διεξάγονται συζητήσει και όπου συνάπτονται δεχομένε συμφωνίε μεταξύ εκπροσώπων κυβερνήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών και είναι πολύ σημαντικέ. Αλλά για να μπορέσουμε να να μπορέσει η Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματικά να δώσει προστιθέμενη αξία, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι διαδικασίες ολοκληρώνονται εγκαίρως και πιστεύουμε ότι αυτό έχει πραγματικά βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Τέλος, κάτι που αναφέρθηκε και είναι ευαίσθητο για τις, ε, τα καυσαέρια των κινητήρων δίζελ. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν τα συνδικάτα. Βέβαια αυτό δεν θα αποτελεί έκπληξη για σας. Συμφωνούμε με την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην συμπεριληφθεί το ζήτημα αυτό στην οδηγία. Βέβαια παραμένει ένα εκρεμές ζήτημα, το γνωρίζω. Όπως σας είπα όμως, σαν εργοδότες εντός Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια, είναι σημαντικό να δούμε εάν συμπερίληψη ουσιών και διαδικασιών στην οδηγία και κάποιες οριακές τιμές αν συμπεριληφθούν, αν αυτό που προβλέπεται μπορεί πραγματικά επιτόπου να εφαρμοστεί. Δεν συμφωνούμε ότι η διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων ε, διζελοκινητήρων είναι κάτι άσχετο, αντιθέτως πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλές μελέτες που έγιναν μέχρι τώρα βασιστήκαν ουσιαστικά σε έκθεση από παλαιούς διζελοκινητήρες και δεν είναι η ίδια κατάσταση που ισχύει με τους νέους ε, διζελοκινητήρες όπου η χημική συγκέντρωση και η σύνθεση των χημικών είναι πολύ διαφορετική. Ό,τι και αν συμβεί στο μέλλον για αυτό το θέμα, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία, και η πρόοδος αυτή επηρεάζει και το επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων. Και πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ ότι αυτή είναι μια περίπτωση όπου ασκούνται πιέσεις από κύκλους της βιομηχανίας. Πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουμε μια τυποποιημένη μέθοδο μετρήσεων στον τομέα αυτό. Βέβαια εξετάζοντας τρόπους ε, βελτίωσης της προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε διάφορες καρκινογόνες ουσίες είναι απίστευτα σημαντικό και συμφωνούμε ως εργοδότες όσον αφορά την προσέγγιση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι γίνεται σε νομοθετική βάση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι αυτό που θεσπίζεται σε νομοθεσία μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί. Ένα παράδειγμα να δώσω. Σε κάποιες περιπτώσεις ξέρουμε ότι εκπομπές από φορτηγά, φερρυπίν, από κινητές δίζελ φορτηγών Ε, λαμβάνουν χώρα όταν στέλνει μια εταιρεία αγαθά με φορτηγό σε άλλη εταιρεία. Και ίσως ο εργοδότης στον τόπο που οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κάποια από τα καυσαέρια από τον διζελοκινητήρα δεν γνωρίζει τι κινητήρα χρησιμοποιεί αυτό το φορτηγό διότι το φορτηγό έρχεται από άλλη εταιρεία. Είναι ένα πρακτικό παράδειγμα όπου δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί η έκθεση σε κάποιες περιστάσεις, κυρίως σύμφωνα με την οδηγία περί καρκινογόνων. Και πρέπει αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη, εξετάζοντας το πώς θα επιφέρουμε βελτιώσεις στις διάφορες οδηγίες. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την άποψη των κοινωνικών εταίρων γιατί πρέπει εμείς οι πολιτικοί να γνωρίζουμε τις απόψεις σας. Αλλά το δεύτερο είναι να έχουμε και τα σωστά επιστημονικά στοιχεία. Οι κοινωνικοί εταίροι και οι επιστήμονες, αυτοί είναι οι συνομιλητές μας. για να καταλήξουμε σε σωστές αποφάσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως πολιτικοί. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε εσείς κυρία Σμιθ. Ότι αν θέλουμε να Πάμε πιο γρήγορα. Μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πολύ καλό αυτό. Αυτό ισχύει και για τους κοινωνικούς εταίρους και για τους πολιτικούς. Βεβαίω θέλουμε να, όταν θέλουμε να δράσουμε πιο γρήγορα, μπορούμε να δράσουμε πιο γρήγορα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρολά, που θα είναι ο εισηγητής μας για αυτή τη δεύτερη δέσμη καρκινογόνο. Αλλά δουλεύουμε ως ομάδα, οπότε συλλογικά θα σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κλοντ, ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές μας. Νομίζω ότι οι παρουσιάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Θα μας επιτρέψουν ε, να καταλάβουμε καλύτερα και να προχωρήσουμε στη δουλειά μας. Και θέλω να χαιρετήσω και την εργασία και το φιλόδοξο χαρακτήρα της εργασίας Κομισιόν. Για το θέμα αυτό Επί μία δεκαετία δεν είχε γίνει τίποτα, τώρα κάτι γίνεται, προχωράνε τα πράγματα, πολλά πράγματα προχωράνε. Χρειαστήκαμε χρόνο για να βάλουμε και πάλι μπρος τη μηχανή, αλλά τώρα αυτή η μηχανή έχει και πάλι πάρει μπρος και ε, θέλουμε και να αναρμονίσουμε αλλά και να βελτιώσουμε την προστασία των εργαζομένων. Αυτή είναι η δεύτερη αναθεώρηση. Ε, μας αναγγέλθηκε και μια τρίτη και ίσως και μια τετάρτη. Αλλά ναι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια μόνιμη διαδικασία αναθεώρηση. Είναι μια διαδικασία που ποτέ δεν θα να σταματάει, γιατί η πραγματικότητα δεν σταματάει. Οι χημικές ενώσει ε, στις οποίες εκτίθενται οι εργαζόμενοι ε, αναπτύσσονται ε, συνέχεια, τροποποιούνται, μπαίνουν καινούργιες. Η εργασία αυτή λοιπόν πρέπει να συνεχιστεί. Ο συζητήτη θα έχουμε την ίδια προσέγγιση όπως κατά την πρώτη δέσμη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι για να προστατεύουμε τους εργαζομένους, αλλά παράλληλα και ρεαλιστές, ούτως ώστε αυτά που προτείνουμε να είναι εφαρμόσιμα. Όπως είπαν διάφοροι, το να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι, χωρίς να έχουμε δυνατότητα εφαρμογής και ελέγχου αυτών που προτείνουμε, δεν έχει έννοια. Το δεύτερο στοιχείο της προσέγγισής μας είναι αυτό που ακούσαμε και τώρα. Πρέπει να βασιστούμε, να ακούσουμε τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και να έχουμε φυσικά και την ε, στοιχειοθετημένη ε, γνώμη των επιστημόνων. Εγώ ως πολιτικός το λέω δεν τις γνωρίζω αυτές τις ουσίες. Για να μπορέσω να προτείνω προόδους στην νομοθεσία πρέπει να έχω τις απόψεις όλων αυτών που γνωρίζουν από κοντά την κατάσταση. Σε ευχαριστώ πραγματικά Μαρίτα και όλους τους ε, σκιώδεις για την πρώτη δέσμη. Χάρη σε όλους σας. Τα πήγαμε πολύ καλά στην πρώτη δέσμη. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί η ίδια καλή απόδοση. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και συνεργαζόμενοι όλοι όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ θα πάρω όλο το χρόνο που χρειάζεται, όχι για να επιβραδύνω την πρόοδο, αλλά για να ακούσω τους εκπροσώπους όλων των φορέων. Και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές επιχειρήσεις, μεγάλες, μικρές, όχι βέβαια για να επιχειρηματολογήσουμε ότι οι εργαζόμενοι στον ε, α τύπο επιχειρήσεων χρειάζονται λιγότερη προστασία, αλλά για να μπορέσουμε να δούμε πώς με βάση τη διαφορετική πραγματικότητα θα επιτύχουμε τους ίδιους στόχους. Νομίζω ότι θα κάνουμε καλή δουλειά για το θέμα αυτό. Βασίζομαι και στους συναδέλφους, βέβαια δεν είναι πάρα πολύ. Αλλά κοιτάξτε, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θα μιμηθώ τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, είναι φυσιολογικό. Αλλά βασίζομαι πολύ στην συνεργασία με τους συναδέλφους μου όπως και πιο συγκεκριμένα στη συνεργασία με τους Κιώδης για να συζητήσουμε τη δεύτερη δέσμη και τις υπόλοιπε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι για να επανέλθουμε όλοι ξεκούραστοι και με ενέργεια για να ασχοληθούμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Κλοντ, βεβαίως και εγώ. Okay. από την Κομισιόν Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δράτω με τις να συγχαρώ και εσάς και τον κύριο Ρολά και τους άλλους βουλευτές για την δουλειά που έκαναν και την επιτυχία ολοκλήρωση. Επίσης, σας ευχαριστώ που κανονίσατε αυτήν την ακρόαση Ευχαριστώ και τους ομιλητές, την ΣΚΟΛ, την Όσα, Αλλά βεβαίως και στο παρασκήνιο γίνεται πάρα πολύ δουλειά για να ετοιμαστούν αυτές οι προτάσεις. Οπότε χαιρόμαστε που είναι εδώ και τους ακούμε και ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. και εύχομαι καλή επιτυχία στον κύριο Ρολάν με αυτή τη το νέο πακέτο και μιλάμε για τρίτο και τέταρτο πακέτο αλλά de facto όπως είπατε κύριε Ρολάν δεν θα τελειώσουν εκεί τα πράγματα θα είναι μια συνεχής διαδικασία. Αλλά μιλάμε για πακέτα, αλλά όπως είπατε είναι κάτι το ρευστό. Μια συνεχής επικαιροποίηση. Να σας ενημερώσω και για κάτι ατύπως. Με λύπησε λίγο το σχόλιο για το lobbying. Και ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την πρόταση της Κομισιόν. Εξ ονόματος της Επιτρόπου τα απορρίπτω αυτά με τα και είναι λυπηρά πραγματικά αυτά τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων. Σας ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Ε, το σχέδιο έκθεση για το δεύτερο πακέτο θα ετοιμαστεί στις 17 Οκτωβρίου, η εξέτασή του 9 Νοεμβρίου, η προθεσμία τροπολογιών 14 Νοεμβρίου και μετά θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τον Ιανουάριο του 2018. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας καλοκαίρι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE